Κάνουμε αυτή την ακρόαση σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας που καλύπτεται από το ψήμα του 2016 για, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει μια διοίκηση ανοιχτή. Σήμερα είναι 28η μέρα της κινητοποίησής μας κατά της μονομερούς επιβολής από τη δίκη του Κοινοβουλίου σκληρών συνδικών εργασίας. Χρειάζεται πολιτική διαμεσολάβηση. Δεν θα επιτρέψουν πέραβαση ωραρίου στι συνεδριάσει. Ευχαριστούμε για την κατανόηση από την πλευρά των διαρμηνίων. Οπότε πρώτα για κάποια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί από κάποια αξιολόγηση κόστου ωφέλου και αιτήσει τη Επιτροπή ε, Γιούρη. Η ε, Υπηρεσία Έρευνα του Κοινοβουλίου πρόκειται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ε, αυτής της μελέτης επιπτώσεων και τα αποτελέσματα της ε, δημοσίας διαβούλευσης για το πώς θα έχουμε ε, ένα διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή τη μελέτη θα αξιολογήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις της πρότασης του Κοινοβουλίου και της ε, διαβούλευσης. Οπότε να έχουμε καλύτερη κατανόηση της εμπειρίας πολιτών αλλά και φορέων όσον αφορά τις συναλλαγές τους με την δίκη της ε, Ένωσης και θα εξολογήσουμε το πώς εφαρμόζονται οι διοικητικές διατάξεις και πώς ε, λειτουργούν οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη μας χαρά να καλωσορίσουμε τον πρώτον την πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερ μας, αλλά και την κυρία Οράιλη, την ε, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Βλέπετε ότι αυτό το θέμα ελκύει ενδιαφέρον και την προσοχή της πολιτικής τάξης στην Ευρώπη. Οπότε θα ακούσουμε τι έχετε να πείτε και θα ακούσουμε και τους εμπειρογνώμονες, τον καθηγητή Χέρβικ Χόπμαν και τον κύριο Ντέρκ Χιούντιχ. Τους ευχαριστώ που ήρθαν και εκείνοι. Τώρα, ευθύ εξ αρχής θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χάουτελα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στην ακρόαση. Έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρονάκια που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια σε αυτή την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η δίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον Ιανουάριο του 2013, πάνω από πέντε χρόνια πριν δηλαδή, ε, εγκρίθηκε αυτό το διοικητικό δίκαιο, το οποίο τώρα ονομάζεται ο κανονισμός για μια διοίκηση στην Ευρώπη που θα είναι αποτελεσματική ε, και ανοιχτή όπως ορίζει η συνθήκη. Και έτσι ε, θέλουμε να κατοχυρεί το δικαίωμα σε μια χρηστή διοίκηση, ε, να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με ασφάλεια δικαίου, χωρίς παραθυράκια. Και όλα αυτά να συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο και να ανταποκρίνονται στο κράτος δικαίου που θέλουμε να πρετανεύει. Πριν από 18 χρόνια, ο Ιάκομ Σόντερμαν, ο πρώτος διαμεσολαβητής, όρισε τις αρχές της χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς που είναι στοιχειώδες για κάθε υπηρεσία, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο κόσμο από αυτή την υπηρεσία. Και ήδη ευκνήσει ότι με αυτή την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πρωτοπόρα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών και να μην είναι ο πόδιο Πομπέο τράγος. Και νομίζω ότι αυτό που είπε τότε, ο κ. Σούτερμαν ισχύει 18 χρόνια μετά. Τώρα κατηγορούμεθα ε, ότι είμαστε η αιτία των που προσπαθούμε να λύσουμε. Και σε πάρα πολλά κράτη-μέλη ε, υπάρχει τέτοια δυσπιστία, κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμαστε, δεν πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό και τώρα θέλουμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση, κάναμε τη δημόσια διαβούλευση και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί ε, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και το Κοινοβούλιο και αυτό το ψήφισμα. Πριν από δύο χρόνια είπε η Επιτροπή ότι το κόστος της κωδικοποίησης του ιδιωτικού δικαίου είναι πιο σημαντικό από τα ωφέλη και σχεδόν κλείθηκε το Κοινοβούλιο να κάνει αυτού του είδους την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της κωδικοποίησης. Ε, αυτό κάναμε. Και θα ακούσουμε σύντομα τα αποτελέσματα. Οι αρχές μιας χρηστής διακυβέρνησης όπως νομιμότητα, αναλογικότητα, προσβασιμότητα στα έγγραφα, ισότητα, αποφυγή δυσμενών διακρίσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να κατευθυντήρω για την ε, ευρωπαϊκή διοίκηση για κάθε απόφαση. Πάντως φοβάμαι ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε και αυτές οι αρχές μπορεί να μην εφαρμόζονται με συνέπεια, να μην εφαρμόζονται καθόλου. Και αυτό οδηγεί σε περιπλοκές διοικητικές. Από ό,τι μου είπαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κάθε φορά που υπάρχει κατηγορία για κακοδιοίκηση, αναλύει την κάθε περίπτωση χωριστά. Αλλά πολλές φορές αυτό που ισχύει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί το ποια είναι κάθε φορά η ορθή διαδικασία, ποια είναι τα διαδικαστικά δικαιώματα κάποιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. Ε, και ε, έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε όλοι να μπορούν να συναλλαγούν με κάποια ανοιχτή, ανεξάρτητη και αποτελεσματική διοίκηση. Και βεβαίως και εμείς έχουμε τον ίδιο στόχο. Η διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε, είναι, ούτε πρέπει να είναι κάτι το στατικό, μια οντότητα αμετάβλητη μέσα σε έναν κόσμο και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μεταβάλλεται συνεχώ. Η ψηφιοποίηση είναι η σημερινή κυριαρχή τάση και η δυνατότητα να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Είμαι πεπισμένη ότι αν έχουμε ε, συνεπή και πλήρη νομοθεσία και διοικητικό δίκαιο θα είναι τα πράγματα πιο εύκολα. Εν τέλει, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρώτον υπρόεδρο της Επιτροπής που ήρθε εδώ. Πάντοτε είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε πώς θα βελτιωθεί η λειτουργία της Ένωσης. Επίσης, ευχαριστώ θερμά την κυρία Οράιλε, την Δημοσιολαβήτρια, γιατί συνεχώς προσπαθεί να προωθήσει αυτές τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας σήμερα. Επίσης και τον κύριο Χόφμαν και τον κύριο Χιούντιχ, οι οποίοι προσφέρουν ε, από λάση πανεπιστημιακών τις πολύτιμες ε, απόψεις τους, και περιμένω πώς και πώς να ακούσω την γνώμη σας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Φραντ Τίμερμαν να πάρει τώρα το λόγο. Πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που με καλέσατε να σας μιλήσω σήμερα. Τον Απρίλιο, όπως άλλωστε τακτικά το πράτο, τοποθετήθηκα στην Επιτροπή σας ε, και δεσμεύτηκα ότι θα μπορούσα να έρθω για την ακρόαση. Άλλωστε επιλογή δεν είχα γιατί με εκλήτευσε η κυρία Χάουταλα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Η Επιτροπή βεβαίω είναι προσλωμένη στην εξασφάλιση για τι επιχειρήσει, του καταναλωτέ, του πολίτε και όλου του εμπλεκόμενου φορεί ενό συστήματο διοικητικού ανεξάρτητου, ε, διαφανού, αποτελεσματικού και πάνω απ' όλα με λογοδοσία. Υπάρχει ένα σύνολο εγκάρσεων κανόνων, όπως και σε κάθε άλλο διοικητικό σώμα, που διέπουν όλη τη λειτουργία, όπως ο κώδικας χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς, ο κώδικας συμπεριφοράς για τους επιτρόπους. Και θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι η αναθεωρημένη του έκδοση ε, τέθησε ισχύ τον Φεβρουάριο, αλλά και τις διατάξεις του κανονισμού προσωπικού, του δημοσιονομικού κανονισμού, πρόσβαση στα έγγραφα και άλλα. είναι σημαντικό οι ρυθμίσει πάντα να επαληθεύονται σε σχέση με κάποιε αλλαγέ που ενδεχομένω να έχουν λάβει χώρα σύν το χρόνο. Συμβαίνει αυτό πάντα. Και πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε και να προσαρμόζουμε την νομοθεσία με τι εξελίξει στη διοίκηση. Να δίνουμε πάντα το καλύτερο παράδειγμα. Για του εγκάρσιου κανόνε και πρακτικές, η καθημερινή δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από τι αρχέ τη χρηστή διοίκηση νομιμότητα, αναλογικότητα, πρόσβαση στο φάκελο, υποχρέωση ε, αιτιολόγησης, ισότιμης μεταχείρισης, μη διακρίσεως, ε, ισότιμης χρήσης των γλωσσών, βεβαίως. Η Επιτροπή αναλύει κάθε περίπτωση και υπενιγμό κακοδιαχείρισης και καταλήγει στα συμπεράσματα που απαιτείται. Επικοδομητικά δεν ανταποκρινόμεθα στα αιτήματα της ε, Ευρωπαίας ε, διαμεσολαβητή η οποία πάντοτε έχει πολύ επικοδομητικό ε, ρόλο και αυτό μας διευκολύνει ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολλές και Διαφορετικέ δραστηριότητε, μια ποικιλία δραστηριοτήτων που υπάρχονται και σε δικού του ειδικού κανόνε όπω τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή τα θέματα του ανταγωνισμού. Και εδώ πέρα υπάρχει ειδική εγγύηση, εγγύηση ειδικών διοικητικών δικαιωμάτων για τους πολίτες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς αυτούς μπορεί να έχουν εκτεταμένες συνέπειες για τους πολίτες αυτούς. Για την ε, δημόσια διαβούλευση σημειώνω 2% των ε, ανταποκριθέντων έχουν θετική αντίληψη, 36% αρνητική για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επίσης, ε, γενική αντίληψη των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δείχνει πολύ θετικά και πολύ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι περίμενε. 75% των ανταποκρινωμένων απαντούν ότι γνωρίζουν τι ίδιους υπηρεσίες προσφέρουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προς το κοινό και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υποστήριξη με 76% εκδηλώνουν οι ανταποκριθέντες ε, στην ε, εισαγωγή επιπλέον μέτρων για την ενίσχυση των διοικητικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα. Στο γιατί θέλουν να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απαντήσεις ήταν με 75% να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και με 50% να βελτιωθεί η διαφάνεια στη διοίκηση Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίω, πάντα παραμένουν ανάμεικτα τα συναισθήματα που εκφράζονται σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία της διοίκησης. Ε, παραδείγματι νέα νομοθεσία με ελάχιστε προδιαγραφέ, νέα νομοθεσία με εναρμόνιση, ε, καλύτερη εφαρμογή τη υφιστάμενη νομοθεσία, τεχνικέ λύσει για την εξασφάλιση, την απλούστευση μάλλον της ε, πρόσβασης, ε, στη διοίκηση, για το κοινό. Όλες αυτέ οι απαντήσει έχουν δοθεί. βεβαίω η Επιτροπή θα εξετάσει και τι απαντήσει αυτές και την, ε, ε, τα πορίσματα τη σημερινή συζήτηση κατά την αξιολόγηση της. Και βεβαίω οι υπηρεσίε μα ακόμα για χρηστή, εγώ να αποχωρήσω, θα, θα κρατήσουν πολύ προσεκτικέ σημειώσει και περιμένουμε. Επίσης, με βάση και επανερχόμενα ζητήματα που επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και προβλήματα, ε, και τι συζητήσει τι σημερινέ να συνδυάσουμε για να βρούμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε στη διαθέση για καλύτερη συνεργασία, ε, πάντα με στόχο τη βελτίωση της ε, ζωής των πολιτών. Θέλω να πω ότι για μένα ταμπού δεν υπάρχουν, θέλω πάντα την καλύτερη λύση, αλλά πρέπει και να με πείσετε. Πράγμα το οποίο, όπω λένε οι συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο πάντα. Η Επιτροπή με πολύ μεγάλη σοβαρότητα επιδιώκει την ε, πίτευξη του στόχου για τον πολίτη μιας ευρωπαϊκής διοίκησης αποτελεσματικής, διαφανούς, ανοιχτής, πάνω απ' όλα όμως με υποχρέωση λογοδοσίας στον κυρίαρχο της, στον κυρίαρχό της που είναι ο Ευρωπαίος πολίτης και οπωσδήποτε έχει και η Ombudsman, η Μεσολαβήτρια, πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ρόλο διαδραματίσει εδώ θέλουμε να έχουμε τα ύψιστα επίπεδα δημόσιας διοίκησης, όπως τα γνωρίζουν χώρες Ευρώπης ή του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να είναι πάντοτε να αναθεωρήσει οτιδήποτε θεωρεί δεδομένο, ότι δεν θα αποκλείσει κάποια ε, σκέψη η προοπτική για αναθεώρηση και με αυτό το πνεύμα έρχομαι να ακούσω τις συζητήσεις, την ακρόασή σας και πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να βρούμε και μια αντίστοιχη στάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα θεσμικά όργανα όλα μαζί θα βρούμε μια καλή και θετική λύση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τιμμαντμάνς. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τατιάνα Έβασε από την ομάδα προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας του EPRS να μας παρουσιάσει την δημόσια διαβούλευση ε, σχετικά με τον νέο διοικητικό ευρωπαϊκό νόμο. Έχετε τον λόγο, κυρία Τατιάνα Έβασα. Καλό απόγευμα σε όλους σας και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω αυτήν την δημόσια διαβούλευση και ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς που δώσατε ήδη κάποια ε, στοιχεία ε, και νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα πλέον να κάνω κάποιες επιπλέον παρουσιάσεις σχετικά με τα στοιχεία. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ σωστό ε, ε, να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, υποστηρίζουν τη δράση, θέλουν δράση δηλαδή, θέλουν να έχουν δράση η οποία θα τους δώσει το δικαίωμα ε, ε, να ε, τους δίνει η διοίκηση σωστές και εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις. Επομένω, καλά με τις συζητήσεις, αλλά αρκεί η συζήτηση. Τώρα χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις. Εγώ πρώτα εν είδη εισαγωγής θα απαντήσω στο γιατί, γιατί αυτή η διαβούλευση και γιατί το θέμα είναι ε, ε, σοβαρό. Και θα ξεκινήσω από αυτό το γιατί, γιατί έτσι είναι καλύτερα να κατανοήσει κανείς ε, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Μετά, στο δεύτερο βήμα, θα δώσω λεπτομέρειες για αυτήν την δημόσια διαβούλευση. Πρώτα απ' όλα αυτό το μεγάλο γιατί, αυτή η ερώτηση. Καινοτομία, η κυρία Χαουτάλα το είπε, δεν θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θέλουμε κοινοτομία, όχι μονάχα στην τεχνολογία και στα μεγάλα πράγματα, θέλουμε ε, καινοτομία και στην ε, διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτή έρχεται σε διάδραση με τους πολίτες. Χρειαζόμαστε επομένως προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και σα εξηγώ γιατί. Πρώτον, ε, γιατί ε, η ε, διακυβέρνηση βασίζεται τα μάλλα στη διοικητική μετερρύθμιση η καθημερινή επαφή και οι συναλλαγές ε, του πολίτη με την διοίκηση, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο πολίτης αυτήν την διοίκηση, ε, δεν αφορά μονάχα τα πολύ μικρά διαδικαστικά στοιχεία, αλλά αφορά την πραγματικότητα, τον τρόπο με τον οποίο ε, ζει την πραγματικότητα αυτή, ζουν την πραγματικότητα αυτή οι πολίτες. Επομένως πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μακρά ιστορία ε, ε, προσπάθειας ε, να πιστούν και να πιεστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, φορείς και ο διαμεσολαβητής έτσι ώστε ο συνήγορο συγγνώμη, έτσι ώστε να προωθηθούν τα θέματα αυτά. Ένα δεύτερο στοιχείο γιατί πρέπει να γίνει δηλαδή αυτή η ανανέωση είναι ότι άλλαξαν οι καιροί πλέον. Αρχικά η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν έτσι μια ολιστική προσέγγιση ε, της ε, ε, διοίκησης, γιατί το επιχείρημα ήταν ότι πρόκειται για έμεση διοίκηση και γι' αυτό λέγαμε μερικοί νόμοι από εδώ, κάποιες άλλες ρυθμίσεις από εκεί, μια σωστή διοικητική συμπεριφορά, αλλά πάντα στα πλαίσια του soft law. Τώρα, τώρα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε άλλωστε με την εργασία μας, λέμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100.000 ε, περιπτώσεις διάδρασης ε, σε καθημερινή βάση ανάμεσα στους πολίτες και τη διοίκηση. Ε, και αυτές δεν είναι οι πιο προηγμένες, ας πούμε, οι προηγμένοι υπολογισμοί. Α, δείχνετε και τις διαφάνειες. Ωραία. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλές περιπτώσεις. Δεύτερον, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κατακαιρματισμένο και περίπλοκο όσο έχει σήμερα. Και τρίτον, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει ανάληψη δράσης. Αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο γιατί και γιατί πρέπει να γίνει ε, ε, και γιατί είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση για την διοίκηση και τη σχέση με τους πολίτες. Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σε μεγαλύτερες ε, λεπτομέρειες. Βλέπετε, βλέπετε γενικές πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έχουμε την ε, δική μας έρευνα ε, βασιζόμενοι και στην προσωπική μας ε, εμπειρία. Και βεβαίως η ε, στόχη της έρευνας είναι να δούμε τις προσωπικές εμπειρίες των πολιτών που έρχονται σε επαφή με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά να δούμε την γενική αντίληψη και τη στάση απέναντι στην διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος ποια θα μπορούσε να είναι η υπεραιτέρω δράση θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεθοδολογικές λεπτομέρειες ε, δίνω βεβαίως ε, ε, στην επίσημη, στα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας. Είναι δημόσια διαβούλευση, έγινε σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρχε μια ανάμιξη πολλαπλών απαντήσεων και ανοιχτών απαντήσεων. Είχαμε 166 πλήρεις απαντήσεις από 20 κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τα ευρήματα, ε, ε, ε, όσον αφορά πρώτα τις εμπειρίες, σε τρεις πόλους λοιπόν έχουμε επικεντρώσει ε, τα ευρήματα. Ε, στην ουσία ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα όσον αφορά την διάδραση ανάμεσα στους πολίτες ε, και τη διοίκηση. Ε, θελήσαμε λοιπόν να μάθουμε πρώτα γιατί και πόσο συχνά οι πολίτες έρχονται σε επαφή με τη διοίκηση η πρόσβαση σε ε, πληροφόρηση και η πρόσβαση σε έγγραφα φαίνεται να είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ένας πολίτης θα έρθει σε επαφή με τις, ε, ε, με τις τα διοικητικά όργανα. Και μετά είναι η επαφή με τον συνήγορο κλπ. Θέλησαμε να μάθουμε όμως και γιατί δεν έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Η πιο συχνή απάντηση είναι ότι δεν χρειάστηκαν κάτι τέτοιο. Ωραία, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά στην επιπλέον αιτιολόγηση 70% ε, των ερωτηθέντων είπαν ότι ακόμα και αν ε, είχα μια ανάγκη δεν θα ήξερα πώς να έρθω σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. 7% ε, είπαν ότι ναι θέλουμε 7% είπαν ότι δεν ξέρουμε καθόλου πώς να έρθουμε σε επαφή. Επίσης, ε, ε, η αξιολόγηση της εμπειρίας ε, είναι πολύ μεικτή. Άλλοι είπαν ότι 24% είπαν ότι είναι αρνητική και από το υπόλοιπο ποσοστό περίπου η μισή είπαν ότι ήταν θετική και οι άλλοι πολύ θετικοί. Εάν δείτε λίγο αυτήν την διαφάνεια, ε, θα δείτε διαφορετικές στάσεις ανάλογα και αντιμετώπιση ανάλογα με, την, με το όργανο. Βλέπετε λοιπόν, ανάλογα με την υπηρεσία, ότι τα ποσοστά διαφέρουν βλέπετε ότι υπάρχουν αρνητικές και πολύ ε, αρνητικές ε, απαντήσεις από 6 μέχρι 26% όσον αφορά το, την έψο. 46% των πολιτών είχαν αρνητική ή πολύ αρνητική εμπειρία. Επίσης, διαφορετική αντιμετώπιση ε, για κάθε, ε, για κάθε ένα όργανο ανάλογα ε, με την διαφορετική εμπειρία που έχουν οι πολίτες. Αν δούμε, μπορούμε να δούμε και μέσους όρους βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις διαφορές ανά υπηρεσία. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα και να δούμε ποια, ποιες είναι οι άλλες θετικές και αρνητικές τάσεις ε, που βασίζεται η θετική ή αρνητική εμπειρία των πολιτών. Βλέπετε στις πρώτες γραμμές ε, ότι ε, ως κύριο πρόβλημα είναι η βραδύτητα των διαδικασιών. Βλέπετε ότι εδώ έχει ένα 42%. Ε, επίσης, ε, η διαδικασία του να βρει κανείς τις, πληροφορίες, τις που θέλει ε, όσον αφορά την προσβασιμότητα και των υπηρεσιών, σε αυτή τη διαφάνεια επίσης το βλέπετε, είπαν πολλοί ότι, θα μπορού, ότι είναι ικανοποιητικός ο βαθμός της προσβασιμότητας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε το κόστος. Εμείς ρωτήσαμε ποιο θεωρούν το μεγαλύτερο πρόσκομα και λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη διαφάνεια είπαν ότι το κόστος της λειτουργικής ασυνέχειας ε, ήταν κατά την άποψή τους το μεγαλύτερο. Εμείς έχουμε δώσει εδώ ε, τέσσερα διαφορετικά είδη κόστους ε, και το πιο σημαντικό ήταν αυτό το operational incoherence cost. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, οι πολίτες ε, υποστηρίζουν την λήψη περαιτέρω δράσης. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, αλλά σε γενικές γραμμές 76% υποστηρίζουν μια τέτοια δράση. Το δεύτερο στοιχείο τώρα που αφορά τη γενική στάση. Θα δείτε λοιπόν εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία Νομίζω ότι τα κεντρικά στοιχεία εδώ είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα 44% εξακολουθούν να θεωρούν δύσκολο ή πολύ δύσκολο να έρθουν σε επαφή ή να πάρουν πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Ε, ανεξάρτητα από όλες τις τεχνικές λύσεις, 44% των πολιτών και των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι δύσκολο ή και πολύ δύσκολο να έρθουν σε επαφή με την διοίκηση. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο προβληματικό κατά την άποψή μου βρίσκεται στα δεξιά πλευρά ε, της διαφάνειας ε, γιατί υπάρχουν πολλές ε, στρεβλές ε, σκέψεις ή αντιλήψεις από πλευράς των πολιτών. Και όσον αφορά τις διαδικασίες και τα δικαιώματά τους, ε, διαπιστώσαμε ότι για τα θέματα αυτά ε, υπάρχει δυσκολία κατανόησης. 52% ε, δεν γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες. 40% όλων των ερωτηθέντων πιστεύουν εσφαλμένα ότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν τους δίνει δικαίωμα πρόσβασης στην διοίκηση. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, ε στρεβλή αντίληψη και ε, σύγχυση όσον αφορά ε, το θέμα αυτό. Θα σας δώσω βέβαια, θα σας αφήσω και τα έγγραφα και το σύνολο της μελέτης έτσι ώστε να τη μελετήσετε κι εσείς σε βάθος. Πάντω εξακολουθούν, όπως λέω, να υπάρχουν θέματα τα οποία προκαλούν σύγχυση στο πνεύμα των πολιτών. Τρίτο στοιχείο της ε, και τμήμα τη παρουσίασής μου, η περαιτέρω δράση, μελλοντικέ δράσεις δηλαδή. Όπως είπα και προηγουμένως, 75% των πολιτών, άρα πολύ ισχυρό τμήμα των πολιτών, ζητούν επιπρόσθετα μέτρα. Ζητήσαμε να μάθουμε ε, ποιες θα ήταν ε, ε, από τους πολίτες, ποιες θα ήταν οι διάφορες δυνατότητες, θα ήταν soft law, αν θα ήταν κανονικός νόμος κλπ. Είναι σαφές ότι προκύπτει τάση 82% των ερωτηθέντων μας είπε ότι ζητούν νομικώς δεσμευτικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα και η διαφάνεια. Στην τελευταία μου διαφάνεια ε, σας μεταφέρω τρία κεντρικά μηνύματα. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν δυσκολίες όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος τους για καλή διοίκηση. Δεύτερον, ότι οι απόψεις τους και οι εμπειρίες τους ε, δεν είναι παρόμοιες ε, και αυτό το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να μας κινήσει την προσοχή είναι ακριβώς η σύγχυση η οποία επικρατεί πέρα τα ε, ευρωπαϊκά διοικητικά θέματα και τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι η υποστήριξη των πολιτών για επιπλέον δράση. Όσον αφορά τώρα την καινοτομία, επανέρχομαι σε αυτό, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κανόνες ε, και πρέπει να βρούμε λύσεις. Και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι νόμοι, από τη στιγμή που υπάρχουν οι διαδικασίες, αυτό που λείπει είναι αυτή η καινοτομία, αυτές οι καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα φέρουν τους πολίτες κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη. Ε, σας... Ε, ε, ε σας ε, παρακινώ λοιπόν να διαβάσετε αυτές τις 70 σελιδούλες της έρευνας έτσι ώστε να δείτε όλα τα στοιχεία αναλυτικά με αριθμούς και λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Λέω Πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή Ανδρέα Ρέντα ο οποίος είναι ε, ερευνητής, ανώτερος ερευνητής στο CPS, e για να σας παρουσιάσει ε, τις επιπτώσεις ενδεχομένων πρωτοβουλίων της Ένωσης. Σας ευχαριστώ κυρία Άουταλα, κυρία Οράιλη, Δημεσολαβήτρια, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, μέλη της Υπηρεσίας Έρευνας του Κοινοβουλίου και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι που είστε εδώ για αυτό το σημαντικό θέμα. Θα παρουσιάσουμε μία μελέτη. Αυτή διεξήχθη από το κέντρο μελετών μας και έχουν συμβάλει και δύο συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπεργκ που παρίστανται και θα μπορέσουν να απαντήσουν ενδεχόμενες ε, ερωτήσεις σας η κυρία Μέγουβες και ο κύριος Κολόμπο. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Μας πήρε κάποιους μήνες αυτή η μελέτη. Επίσης όμως έχουμε βασιστεί σε έρευνες προηγούμενες και του Κοινοβουλίου, του, στις υπηρεσίες ερευνών και πανεπιστημίων και κάποιων think tanks που έχουμε εδώ εκπροσώπους τους σήμερα. Το Risk Forum Επίσης που έχουμε εδώ εκπρόσωπο και όλα αυτά μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε τα επιχειρηματά μας όσον αφορά τις επιπτώσεις για εναλλακτικέ πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Επομένως, η μεθοδολογία αυτής της αξιολόγησης είναι σύντονη με τις καυτήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για καλύτερη νομοθεσία. Και προσπαθήσαμε έτσι να αξιολογήσουμε το πόσο θα ωφελούσαν κάποιες εναλλακτικέ λύσεις για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση. Επίσης, με μεγάλη μου χαρά, εφήρμοσα τη σχετική μεθοδολογία γιατί έχω και εγώ συμβάλει με μία μου μελέτη το 2013 στη διαμόρφωση αυτών των κατευθυντηρίων. Όταν θέλει κανείς να περιχαρακώσει κάτι το οποίο είναι κατετμημένο θα πρέπει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ, κάτι το οποίο προκύπτει από αυτή τη διαφάνεια χρειάζεται έρευνα και εργαστηριακή ούτως υπήν στο γραφείο και ε, στον πραγματικό κόσμο. Οπότε συνεργαστήκαμε με την Μεσολαβήτρια, εγώ και ο κύριος Κολόμπο. Ε, κοιτάξαμε τι καταγγελίες μου γίνει, τι παράπονα και κυρίως συλληφθήκαμε με την ε, Επιτροπή και Εποχή Γιούγκερ. Λάβαμε υπόψη τους κώδικες ε, ορθής ε, συμπεριφοράς ε, όπως προβλέπονται για τα διάφορα όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συγκεράσουμε αυτά τα αποτελέσματα για να κάνουμε μια καταγραφή του τι καλύπτεται από αυτούς τους κώδικες που διεύγουν το διευθυνό όργανο. Και κάναμε επίσης και κάποια εργαστήρια με πανεπιστημιακούς, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε, σε όλη αυτή την έρευνα αναλύσαμε τα αποτελέσματα ε, της ε, διαβουλεύσης, όπως είπε η Τατιάνα προηγουμένως. Να δούμε επομένως τι μπορεί να αποτιμηθεί ποσοτικά γιατί δεν μπορεί να αποτιμηθεί ποσοτικά από τη φύση του. Όπως ας πούμε η υποχρέωση λογοδοσίας, η νομιμότητα. Δεν είναι εύκολο αυτά να υπολογιστούν. Άλλες όμως μεταβλητές επιδέχονται μια τέτοια ποσοτική ανάλυση. Οπότε στο τέλος θα δείτε ένα πίνακα αποτελεσμάτων με τέτοιους υπολογισμούς. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα χάραξης πολιτικής. Βλέπετε εδώ τώρα αυτόν τον ας πούμε χάρτη. Προσπαθήσαμε τα πράγματα να είναι όσο γίνεται πιο εύκολο να αποτυπωθούν, να είναι όσο γίνεται πιο άμεσα. Εδώ αναφέρουμε διάφορες υπηρεσίες, θεσμικά όργανα και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κάποιον ε, κώδικα ορθής ε, συμπεριφοράς και χρηστής ε, διοίκησης. Στη συνέχεια του κώδικα του 2001 του Ευρωπαίου Διεμεσολαβητή. ως επομένως όσες υπηρεσίες ε, υιοθέτησαν και χρησιμοποιούν αυτόν τον κωδικό. Κάποιες υπηρεσίες έχουν το δικό τους όμως κώδικα. Βλέπετε επομένως άσπρο χρώμα μπλε χρώμα και γαλάζιο χρώμα όσοι παραπέμπουν στον κώδικα. Έχουμε την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου και μελετήσει με αυτούς τους ε, κώδικες να δούμε τι διατάξεις ε, καλύπτονται και ποιες διατάξεις δεν καλύπτονται. Στο μπλε βλέπετε την αποτύπωση του πόσο οριακά είναι κάποια πράγματα όσον αφορά το, επίσης το πόσο κοντά φτάνουν αυτοί οι κώδικες σε ό,τι έχει ορίσει το Κοινοβουλίο. Μετά από τις 12 η ώρα ας πούμε στο ρολόι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που δεν καλύπτονται καθόλου όπως ας πούμε το δικαίωμα εκπροσώπησης από συνήγορο, το δικαίωμα για επιβάρυνση οικονομική λογική, ε, το δικαίωμα επικοινωνίας από απόσταση ή ιντερνετικά, την διόρθωση κάποιων ε, λαθών, την υποχρέωση συνεργασίας, όλα αυτά συνδέονται κατά κάποιο τρόπο έμεσα ή όχι τόσο πολύ από αυτούς τους κώδικες παραπέρα, βλέπετε το που το καλύτερα. Ε, σύγκρουση συμφερόντων, προσβασιμότητα σε φάκελο, υποχρέωση τήρησης ε, αρχείο συμμόρφωσης με νόμο προστασίας δεδομένων και τήρηση χρονοδιαγράμματος και προθεσμιών. Όλα αυτά βλέπετε καλύπτουν ή καλύπτονται από τους υπάρχοντες κώδικες. Το θέμα τι γίνεται από τις 65 αυτές υπηρεσίες σε 35 δεν υπάρχει κώδικας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες, γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, καταστατικά, κανονισμός προσωπικού, αλλά δεν υπάρχει επίσημα κώδικας. Άρα ε, πιο δύσκολο κανείς να δει τι ισχύει από πλευράς διοικητικής διαδικασίας και σχέσεων με το κοινό. Στην επόμενο, τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε αυτούς του τις 65 υπηρεσίες και εδώ έχουμε δύο επιλογές. Στο πράσινο βλέπετε ε, τι γίνεται με αυτή που ήταν πριν, με τις υπηρεσίες που ήταν ε, στο σκούρο μπλε, δηλαδή που έχουν έναν κώδικα. Μετά βλέπετε κάποια λιγότερο συντηρητική πολιτική. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που έχουν θεσπιστεί και μην υπάρχει κώδικας. Είναι αυτό το ανοιχτό πράσινο. Εδώ καλύπτονται αυτές οι λιγότερο συντηρητικές επιλογές. Βλέπετε εδώ να καλύπτονται λιγότερες υπηρεσίες. Οι ίδιες διατάξεις, αλλά και στην πιο αισιόδοξη κατάσταση ε, όσον αφορά τους χρονικούς περιορισμούς ή τις προθεσμίες καλύπτονται μόνο οι μισοί οργανισμοί και υπηρεσίες. Οπότε από πλευράς του κοινού δεν μπορεί κανείς να ξέρει 100% τι ισχύει, τι διέπεται αυτούς τους κανόνες. Δεν είναι σαφές. Πότε υπάρχει προβληψιμότητα, ε, πρόσβασιμότητα στις πληροφορίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για εύρεθμη διοίκηση, για να υπάρχει επομένως ε, μια διοίκηση που είναι υπόλογη στο κοινό. Για να δούμε Τώρα στην επόμενη διαφάνεια έχουμε τις διατάξεις που στους ε, κώδικες που υπάρχουν εκεί που μας δώσαν απαντήσεις στην έρευνα οι οργανισμοί έχουμε 100% κάλυψη για κανόνες αρχή, αρχείων και σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Όμως αν προχωρήσετε προς τα κάτω βλέπουμε ότι τα πράγματα ε, είναι το ίδιο όπως ε, ε να υπενθυμίσουν στο κοινό, να μην ε, αυτοενοχοποιείται ε, την αιτιολόγηση σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ. Και τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα. Οπότε όλα αυτά που βλέπω είναι κάτι σαν στιγμιότυπα από ένα σύνολο διαπιστώσεων, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να σας πούμε όλα όσα βρήκαμε με την μελέτη. Θα δείτε επομένως ότι αυτά επανέρχονται και έχουν κατετμημένη φύση. Όλα αυτά προέκυψαν από την διαβούλευση και την συνάντηση όλων των ε, εμπλεκομένων. Άρα, έχουμε ένα τέτοιο σχήμα που κατατείνει στην κατάτμιση και στην ετερογένεια των πρακτικών. Να δούμε τώρα. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Δημοσιολαβήτρια, να δούμε τι ε, παράπονα, τι καταγγελίες έχει λάβει. Βλέπετε εδώ το 2016 και 2017. Τι καταγγελίες έγιναν και το αναλύουμε την αιτία των καταγγελιών. Να δούμε εδώ τι περιπτώσεις κακοδίκησης καλύπτονται. Το 20% το μπλε. Η μπλε αυτή φέτα είναι θέματα διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδεσίας. Προσβασιμότητα σε έγγραφα, στο φάκελο, όλα αυτά ήδη διέπονται από ρύθμιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ήταν ότι μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις παρόλα αυτά και στη συνάντηση οι συμμετέχοντες καθηγητές τα διευκρίνησαν αυτά. Πιο κάτω τώρα. Ε, πορτοκαλί είναι καλή διαχείριση του προσωπικού της Ένωσης. Μετά έχουμε τα πολιτιστικά. Μετά έχουμε την χρηματοοικονομική διαχείριση κλπ. Βλέπουμε επομένως ότι αυτά τα παραπονιακοδιοίκηση επανέρχονται. Ε, πάμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. And, uh, this led us formulate Εδώ βλέπουμε ποια είναι η λογική της παρέμβασης και οι στόχοι. Ε, έχουμε την κατάδυμση της διαδικασίας, βασικά τρία τα προβλήματα, ότι αδυνατίζει το δικαίωμα για την χρηστή διακυβέρνηση, δεν υπάρχει ανοιχτό πνεύμα διαφάνεια και τα θέματα της ε, αποτελεσματικότητας και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς του κοινού. Άρα έτσι ε, αποδυναμώνεται η νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οπότε έτσι και καταλήξαμε στο πιο είναι γενικός στόχος. Επιπίας βάσεως δηλαδή κάτσαμε να συγκρίνουμε τις εναλλακτικέ. Βλέπουμε τώρα πίσω-πίσω μία διαφάνεια, εδώ τα πράσινα κουτάκια. Γενικός στόχος, το πώς θα προωθηθεί, ποιότητα στη διοίκηση και συγκεκριμένο στόχος, το πώς θα ισχύει το δικαίωμα σε εύρυθμη διοίκηση και με τι εγγύησεις θα περιβάλλεται και έχοντας επίσης καλή σχέση κόστο-αποτελεσμα. Τώρα, να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ. Βρήκαμε τρει τέτοιε εναλλακτικέ επιλογέ. Επόμενη διαφάνεια. Μια υποχρεωτική, βασική επιλογή. Τι θα συμβεί εάν δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν κάνουμε τίποτα. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, δεν θα μείνει βέβαια που είναι τώρα. Παρακάτω τώρα είναι η πρώτη εναλλακτική η μηδενική επιλογή είναι το κλασικό για τέτοιε έρευνε, το να μην κάνει κανείς τίποτα. Οπότε η πρώτη εναλλακτική είναι να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα ο κώδικας χρηστής συμπεριφοράς του διαμεσολαβητή. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα πρέπει ο κώδικας να γίνει μία σειρά μέτρων εκτελεστών και δεσμευτικών. Δεύτερη επιλογή, κανονισμός που να διέπει την διοικητική διαδικασία και τη σχέση με το κοινό των θεσμικών οργάνων. Έχουμε βέβαια και άλλες εναλλακτικέ. Για να σας ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Δεν λάβαμε υπόψη για την έρευνα πέραν της δεύτερης επιλογής αυτό που λέγεται maximum εναρμόνιση. Άρα αυτές οι επιλογές για τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες σημαίνουν το ότι θα μπορούν να προσθέσουν κανόνες ή να παρεκκλίνουν από τους κανόνες που υπάρχουν, να αποκτήσουν ευελιξία. Ας πούμε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ΚΟΜΠ, θέλει να έχει έλεγχο των καρτέλ, δύναμη του άρθρου 101. Δεν θα υπόκειται στον κανόνα του να προειδοποιεί τα, τα καρτέλ εκ των προτέρων. Απευθείας έλεγχος. Αλλιώς θα ήταν αναποτελεσματικό το μέτρο. Άρα, λάβαμε υπόψη τέτοιου είδους επιλογές. Ούτε πήγαμε παραπέρα όσον αφορά μια πλήρη διαδικασία όσον αφορά το περιθώριο ελιγμών στην νομοθεσία, γιατί το Risk ε, Forum το πρεσβεύει αυτό. Άρα δεν αποκλείουμε οι εναλλακτικέ να ωφελήσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον, μακροπρόθεσμα. Για να δούμε τώρα μια-δυο άλλες ε, διαφάνειες για την ε, ποσοτική αξιολόγηση του τι μπορεί να γίνει. Αυτό ήταν ε, τολμηρή ενέργεια γιατί το πρόβλημα δεν είναι και τόσο ποσοτικά αξιολογήσιμο. Καταλήξαμε σε κάποια νούμερα που δεν είχαν καταφέρει να τα βρουν άλλες μελέτες. Έχουμε εδώ κάποιες, ε, κάποια, καμπανάκια κινδύνου και θα πρέπει να δούμε το ότι η μηδενική επιλογή δεν ε, αλλάζει τα πράγματα από πλευράς δαπανών, κόστους και το επιπλέον κόστος της πρώτης επιλογής θα ήταν πρώτα πρώτα ας η πρόσβαση σε έγγραφα παραπέρα το να υπάρχει ένα website για αυτό το σκοπό μετά η δήλωση σκοπού και μέτρων το δικαίωμα του να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα εργασίας της Ένωσης και αυτό με επίσης όσον αφορά τις προθεσμίες και εδώ έχουμε κάνει κάποιους υπολογισμούς ε, οπότε καταλήξαμε σε αιτήσιο κόστος 4.700.000 περίπου και 5.988 για τη δεύτερη επιλογή που είναι πιο τολμηρή και άρα οδηγεί σε περισσότερο έξοδο. Να δούμε τώρα παρακάτω. Να δούμε τώρα τι εξοικονόμηση δαπανών υπάρχει. Έχουμε για την πρώτη επιλογή δύο στήλες και άλλες δύο για τη δεύτερη επιλογή. Η πρώτη στήλη αφορά πολίτες, ε, φυσικά πρόσωπα, κατόπιν έχουμε εξοικονόμηση δαπανών από νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις τέλος πάντων για να δούμε τι εξοικονομίες θα υπάρχει για μια σειρά δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από το κοινό σε σχέση με την διοίκηση, εξοικείωση, με την υποχρέωση υπαρχής πληροφοριών, συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία ε, των απαιτουμένων πληροφοριών, συμπλήρωση εντύπων κλπ. Εδώ βλέπουμε αυτόν τον πίνακα για αυτές τις δραστηριότητε που με αυτές τις δύο εναλλακτικέ θα γίνουν πιο απλές. Και επίσης θα εξοικονομηθεί και χρόνος υπολογίζουμε. Οπότε κάναμε αυτό τον χρόνο, ε, τον, ε, κάναμε ώρες και λεπτά και ώρες και καταλήξαμε σε αυτή την εκτίμηση. Είναι πιο πολύ, πιο πολύ ο χρόνος ε, στην δεύτερη επιλογή και κάπως λιγότερος ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί στην πρώτη οψιόν, στην πρώτη επιλογή. Και παραπέρα ότι τι εξοικονόμηση θα υπάρχει αν ε, οι χρονικοί περιορισμοί τηρούνται και εδώ πέρα καταλήξαμε στο ίδιο νούμερο και για τις δύο εναλλακτικέ. Οπότε ε, δεν απέχουμε πάρα πολύ από το σύνολο των δαπανών που εξοικονομούνται και στις δύο επιλογές. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη που αξιολογούνται όπως είπαμε στην αρχή εδώ έχουμε μόνο ένα κομμάτι του ωφέλους γιατί υπάρχουν και άλλα ωφέλη που δεν εκτιμώνται, δεν αποτιμώνται ποσοτικά. Οπότε ακόμα και αν δούμε μόνο την ποσοτική αξιολόγηση ε, βλέπουμε ότι το καλό ε, που θα προκύψει καλύτερο από το κόστος τη δαπάνη που απαιτείται. Οπότε τώρα για να δούμε την ανάλυση κόστους οφέλους. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα χρώματα και όσο πιο έντονο το χρώμα πιο μεγάλο το όφελος. Εδώ βλέπουμε την ανάλυση όσον αφορά την επιβάρυνση τη διοικητική, αν ε, επιλογή. Βέβαια κοστίζει το να γίνουν κατευθυντήριες ε, νόμος δεσμευτικός, ανεβαίνουν τα, οφείλη, τα ωφέλη στη δεύτερη επιλογή και γενικώ. Και όχι μόνο για τα δύο πρώτα θέματα, αλλά όσο πάμε προς τα κάτω, έχουμε και ποιοτική αποτίμηση για την ασφαλεία δικαίου, προβλεψιμότητα κλπ. Και καταλήγουμε και στην αποτελεσματικότητα. Και επίσης λέμε ότι αναβαθμίζεται η προστασία των δικαιωμάτων, η εμπιστοσύνη και η νομοποίηση των θεσμικών οργάνων και δύο τελευταία, δεν ξέρω αν ε, ο καθηγητής Χόφμαν θα μας τα πει καλύτερα, το ότι είναι πιο συμβατά τα ευρωπαϊκά θέματα με το εθνικό διοικητικό δίκαιο και για να σταθούμε στο τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό βλέπουμε εδώ ότι πρόκειψε και από το εργαστήριο με του ότι η Ένωση πάει προς περισσότερη ψηφιοποίηση της διοίκησης και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτή η τάση θα οδηγήσει σε περισσότερες εξοικονομήσεις. Εάν όμως πρώτα είναι προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει streamlining της διοικητικής διαδικασίας, τότε θα υπάρξει ομοιογένεια στο πώς συνεργούν διοικητικά όλα τα θεσμικά όργανα. Όλοι το ίδιο one-stop shop, όλοι τις ίδιες διαδικασίες κλπ. κλπ. Εάν συνεχίσει η κατάτμιση διαδικασιών, δεν θα ωφελήσει για πολύ ψηφιοποίηση. Άρα, εδώ προσθέσαμε στα ωφέλη την ετοιμότητα για να ωφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Α, έχω και άλλε διαφάνειε εδώ στον πρώτα συμπεράσματα. Για να δούμε τώρα τι άλλοι δείκτε, τι άλλα κριτήρια υπάρχουν. Για να τα δούμε εντάχει όσον αφορά την καταγραφή τη αξιολόγηση σε σχέση με το πώς μπορεί να τεθεί σε ισχύ αυτός ο οικονομισμό και πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δει κατά πόσο βελτιώνεται η κατάσταση για την προστασία του δικαιώματα στη χρηστή ε, διοίκηση. Σας ευχαριστούμε και να σας απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις και ελπίζουμε ότι με αυτή τη μελέτη έχουμε βάλει ένα λιθαράκι και κάπως συμβάλαμε στο αξιόλογο έργο σας και για συγκεκριμένα στα όσα έχει κάνει η συγγήτρια Χάουταλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης ε, παρεμβάσεις και αντιδράσεις με τον κύριο Πασκάλη Αρντινή πρώτα. Όχι, από την κυρία Εμίλη Ουράιλη, την ε, συνήγορο του πολίτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Χάουταλα και πιο πριν και με τον ε, πρώτο πρόεδρο Τίμερμαν στα τελευταία 17 χρόνια από την υιοθέτηση από το πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Κώδικα Χρηστή Διοικητική Συμπεριφορά που καταρτίστηκε στην υπηρεσία μου το 2001 έχει διευρύνει τις δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμβαθύνει και, τις έχει, και έχουν γίνει και πιο περίπλοκες οι διοικητικέ δομές τη. Έτσι λοιπόν ε, αναπτύσσομενε ε, και οι τεχνολογίες μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μετατρέψει την ε, σχέση μεταξύ του πολίτη και της διοίκησης και βέβαια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βλέπουμε και από την αξιολόγηση που έχει γίνει πρόσφατα. Ε, ταυτόχρονα η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό καταγράφει ένα στιγμιότυπο με διάφορες διακυμάνσεις με βάση τις προδιαγραφές. Άλλος ε, κάνει αντιπαραβολή με τον ε, κώδικα του 2001, αλλού δεν υπάρχει καν διοικητικός κώδικας και το καθεξής. Εάν τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν αυτή τη στάση, αντιλαμβάνεται νομίζω κανείς πόσο μπορεί να ε, μπερδεύεται ο Ευρωπαίος πολίτης ως προς το τι μπορεί να περιμένει και τι μπορεί να νοείται ως χρηστή διοικητική πρακτική υπό τον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Μπορούμε βεβαίως να κατονομάσουμε τα επιμέρους, επιμέρους σημεία του, του συνόλου αυτού που συνιστά την χρηστή διοικητική πρακτική. Αλλά νομίζω ότι είναι απλά. Ε, ο πολίτης θα έλεγε όταν έρθω να σας βρω προσφέρετε μου μια αποτελεσματική υπηρεσία και αν έχω κάποιο πρόβλημα ακούστε με και προσπαθήστε με βοηθήστε να λύσω το πρόβλημα κατά τρόπο δίκαιο και ταχύ. Ε, ένα μέτρο λοιπόν το οποίο μπορεί να βοηθήσει ώστε να γίνει η δημόσια διοίκηση και απλή και κατανοητή στον πολίτη είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει δηλαδή να ε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι μόνο για να καθισχάσουμε τον πολίτη και να μην ε, προξενούμε δυσφορία, αλλά για να λειτουργεί καλά η διοίκηση σε ένα διοικητικό περιβάλλον περίπλοκο. Πολλέ φορέ δεν υπάρχει σαφήνεια για το τι ακριβώ πρέπει να γίνει, πώ μπορεί να το μετωπιστεί ο πολίτη. Και αυτό οπωσδήποτε έχει τη σημασία του. Αναμφίβολα, η συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων λειτουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστήριζε ένα τέτοιο σύστημα. Ε, τώρα, ο πολίτης, ανάλογα με, το, με ποια υπηρεσία έρχεται αντιμέτωπος, βρίσκει διαφορετικό σύνολο κανόνων, πρακτικών ή ακόμα και απουσία πρακτικών. Ένα ενιαίο διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελήψη ειδικών κανόνων, θα μπορούσε να υπηρετήσει ως ένα γενικό διοικητικό δίκαιο και έτσι μετά να δώσει το χώρο για την ανάπτυξη των επιμέρους διοικητικών ε, διατάξεων. Εγώ βεβαίως ε, ε, ως εκ του λειτουργήματός μου έχω να κάνω περισσότερο με ενδοτικό δίκαιο. Πολλές φορές γίνονται, υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν καταλήγουν σε προσφυγές στην υπηρεσία μου ή κάποιες άλλες μπορούν να αντιμετωπιστούν αλλά με ήπιους τρόπους. η κυρία προσθέμενη αξία ε, που μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία, μια υπηρεσία όπως η δική μου είναι ακριβώς ε, να βοηθήσει τη βελτίωση των ε, σχέσεων και σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα διακριτική ευχαίρεια σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση που μπορεί να προκύψει. Το ότι μια πράξη διοικητική είναι νόμιμη δεν σημαίνει ότι δεν είναι ανήθικη ή ότι δεν απογοήτευσε νόμιμες προσδοκίες ή ότι δεν ε, εξαπάτησε τον πολίτη. Έτσι λοιπόν, ή τις προσδοκίες του πολίτη. Αυτό λοιπόν ε, πρέπει να προσέξουμε ώστε το ευρωπαϊκό διοικητικό περιβάλλον να μην ε, είναι ξένο προς τον πολίτη. Πρέπει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία στον πολίτη με λεπτομερείς κανόνες που θα ε, που δεν θα περιορίζουν όμως το σύστημα προσφυγών και αποκατάσταση των δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Frontex έχουν κληθεί από την υπηρεσία μου επανειλημμένως για θέσπιση διοικητικών μηχανισμών. Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει προειδοποίησεις. Έχουμε υπογραμμίσει τους κανόνες τους σχετικούς με τη σύγκρουση συμφερόντων. Όλα αυτά δείχνουν ότι αν δεν υπάρχουν κανόνες χρειάζεται μερικές φορές η υπηρεσία του συνηγόρου του πολίτη να παρεμβαίνει. Ε, Βεβαίω ταυτόχρονα σημειώνουμε την ακαιρεότητα, την αφοσίωση και την ανθρωπιά με την οποία κάνουν τη δουλειά τους οι δημόσιοι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Ο κώδικας ε, στόχο έχει ακριβώς να προαγάγει τις προσπάθειες αυτές ε, μέσω των βέλτιστων πρακτικών για μια νοοτροπία παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τα ευρωπαϊκά όργανα που θα απευθύνεται στον πολίτη, που θα έχει σε αγνώμονα τον πολίτη. Ένας κανονισμό ε, καλογραμμένο, νομοτεχνικά οπωσδήποτε μπορεί να βοηθήσει στο στόχο αυτό. Ταυτόχρονα όμω αν είναι πολύ ε, στεγνός και πολύ στιγνός μάλλον και ε, σκληρός μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Έχουμε ένα σύστημα κατακαιρματισμένο, το είπαμε. Ο κώδικα του 2001, δουλειά του Κοινοβουλίου, δουλειά τη δική μου υπηρεσία, τη Επιτροπή, άλλων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο διοικητικών προδιαγραφών, χωρί όμω να, να, να βάλουν τέρμα στον κατακαιρματισμό ε, και τη σαραμοποίηση. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα σύνολο κανόνων. Πάντα πρέπει να υπάρχει βέβαια ισορροπία, γιατί και τα όργανα πρέπει να αναγνωρίσουν την σημασία ενό τέτοιου δικαίου και να αντιληφθούν ότι δεν κινδυνεύει η αποτελεσματικότητα και το έργο τους και ταυτόχρονα και ο πολίτης πρέπει να δει ότι υπάρχει σεβασμός των θεμελιωδών του δικαιωμάτων και πάνω απ' όλα αυτού σε χρηστή διοίκηση. Χρειάζεται επίσης ε, να εισαχθούν, ε, να γίνει αντιληπτό ότι οι ύψιστε διοικητικέ προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτάσει επίπεδο άνευ προηγουμένου. Ε, ένα σύνολο κανόνων και αρχών βέλτιστων πρακτικών θα είναι πολύ πιο ε, αποτελεσματικό και θα γίνει ακόμη περισσότερο αποδεκτό, καθώς θα αποτελεί και καλό παράδειγμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αλλά και όλο τον κόσμο. Οι αρχές ε, της διοίκησης του διοικητικού δικαίου είναι πόρος, εκδρώνουν κάνευ για κάθε αρχή προστασίας του πολίτη, που άλλωστε ξέρω ότι υποστηρίζουν και οι συνάδελφοί μου οι εθνικοί συνήγοροι του πολίτη. Υπάρχουν ήδη πολλά κράτη που έχουν ε, ε, γενικό δίκαιο για τις διοικητικές διαδικασίες. Οπωσδήποτε μια τέτοια πρακτική μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα, λοιπόν, να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο χάρτης με την προστασία στο άρθρο 8 των προσωπικών δεδομένων και στο άρθρο 42 της πρόσβασης του δικαιώματος προς τα έγγραφα έχουν βρει έκφραση στον κανονισμό 1049 του 1 και τον 1027 του 1 επίσης, ε, δύο κανονισμούς λοιπόν που καταγράφουν τα λεπτομερέστερα στοιχεία τους. Οπωσδήποτε μπορεί και το άρθρο 41 να μεταφραστεί σε νομοθέτημα με τη μορφή κανονισμού. Κάθε νέο νομοθέτημα, ωστόσο, θα πρέπει να εστιάζεται στις κύριε αρχέ τη βέλτιστη διοικητικής πρακτική, να προσφέρει καλέ υπηρεσίε, καλή πρακτική, να στηρίζεται σε διατάξει που θα επιτρέπουν ε, την την υλοποίηση των στόχων της αποτελεσματικότητας, της δικαιοσύνης, της ισότιμης μεταχείρισης. Οπωσδήποτε εγώ συνεχίζω να εφαρμόζω τους κανόνες που υπάρχουν για τη βέλτιστη διοικητική πρακτική, όπως καταγράφονται στην ομολογία, όπως καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα, Πάντοτε θα προσφέρω την πρακτική μου βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, όπως ε, με τον πρακτικό οδηγό, τον ε, μπορείς ή δεν μπορείς να το κάνεις, ε, do's and don'ts που εισαγάγαμε πέρυσι. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι αυτός ο κανονισμός, αυτή, αυτός ο οδηγός μάλλον, το εγχειρίδιο έχει πλέον καταστεί εγχειρίδιο ε, ενημέρωσης για κάθε νέο προσλαμβανόμενο υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ικανοποιεί επίση το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με, μου προσφέρει ιδιαίτερη στήριξη στην, ε, στο έργο μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον καθηγητή Χοφμάνα, ο οποίος ε, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου για 10 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση σε αυτήν την ακρόαση, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να εξακολουθήσει το Κοινοβούλιο να πιέζει, όπως είπε και η κυρία Χαουτάλα προηγουμένως, με τον ίδιο ρυθμό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση των πραγμάτων, το status quo το οποίο εξετάζουμε είναι συγκεκριμένο τα ίδια προβλήματα ε, ή μάλλον λύσεις τα ίδια προβλήματα μέσω νέων πολιτικών ε, ε, με τρόπο διαφορετικό πολύ συχνά ανεξάρτητα από το κατά πόσον η διαφορά χρειάζεται ή όχι επίσης μεγάλη περιπλοκότητα άνευ λόγου και ελλείψεις, ελλείψεις που δυστυχώς προκύπτουν από το γεγονός ότι αυτές οι ε, ε, συγκεκριμένες προσεγγίσεις των προβλημάτων μονάχα εν μέρη αντιμετωπίζουν το, τα ζητήματα. Χρειαζόμαστε γενικότερες ε, αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ας πούμε το δικαίωμα ακρόασης και αναφοράς είναι διασφαλισμένο ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα. Επομένως δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν οι πολίτες ποια ακριβώς δικαιώματα έχουν έστω αν αυτά υπάρχουν κάπου στον νόμο. Αυτά τα, ε, αυτά τα κενά λοιπόν δημιουργούν πρόβλημα στην εξέλιξη όπως ε, άλλωστε ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως και από αυτήν ακριβώς την κατάσταση προκύπτει σύγχυση στους πολίτες και ασάφεια όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες. Ο Ανδρέα Ρέντα είπε προηγουμένω ε, και ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση δεν είναι μια διοίκηση που παίρνει αποφάσεις όσον αφορά κρατικές επιδοτήσεις ή όσον αφορά τον ανταγωνισμό κλπ. Ε, υπάρχουν πολλές ε, περιοχές και κλάδοι πολιτικής, παιδεία πολιτικής, τα οποία απαιτούν συν αποφάσεις και συν διοίκηση σε εθνικό και νοσιακό επίπεδο αλλά ε, ακριβώς ε, λησμονάται, ε, λησμονείται συγγνώμη, αυτή αυτό το, το ευρύ πεδίο των διτών διοικητικών θεμάτων. Αυτές οι σύνθετες διαδικασίες πολύ συχνά φτάνουν στη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως ας πούμε Best και δεν πρέπει να λησμονούμε την κατάσταση και η πρόταση ακριβώς του, του ε, Κοινοβουλίου για ε, ρύθμιση ε, μας οθεί στο να λάβουμε υπόψη μας τα θέματα αυτά. Υπάρχει κάτι το οποίο διαπιστώνουμε βλέποντας την εμπειρία των κρατών, γιατί είναι δύο τρίτα των χωρών που έχουν ειδικές διοικητικές διαδικασίες, ε, και άλλωστε οι χώρες είναι πραγματικά εκολαπτήρια, εργαστήρια ε, νομικά ε, και νομοθετικών ρυθμίσεων. Διαπιστώνουμε λοιπόν έλεγα ότι προφανώς δεν χρειάζεται να επανεφαεύρουμε τον τροχό γιατί έχουμε Έχουμε χώρες όπως η Αυστρία από το 1925 και η Γαλλία από το 2016 που έχουν κωδικοποιήσει ε, τον ε, διοικητικό τους ε, ε, ε, κώδικα ε, και βλέπουμε ότι και η Πολωνία ας πούμε σιγά σιγά ξεπερνάει αυτό τον πολύ βαρύ εκτελεστικό μηχανισμό των πολλών ετών έτσι ώστε δειλά να ξεκινήσει μια κωδικοποίηση Επομένως ε, πρέπει να δείξουμε ορθολογισμό, πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό ε, και να προχωρήσουμε ε, στις διαδικασίες κωδικοποίησης. Όσον αφορά την διαδικασία μετά την κωδικοποίηση, μπορεί κανείς να δει και την, την μελέτη επιπτώσεων και την αξιολόγηση επιπτώσεων του Κοινοβουλίου. Από την άλλη πλευρά, η Administrative Procedure Act ε, μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά στην ουσία ε, αποτελεί ε, μια παρένεση για απλούστευση, αλλά η απλούστευση είναι πάντα μεγάλη πρόκληση ε, για την Κομισιόν και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν δει κανεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μπουν σε μια γενική συμφωνία, ε, πράγμα αρκετά απλό να γίνει, θα διαπιστώσουμε ότι αποτελεί ακριβώς αυτή η κίνηση ένα πάρα πολύ μεγάλο πρώτο μεγάλο βήμα και η πρόταση κανονισμού του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ακριβώς μια συνεκτική αντιμετώπιση του θέματος των διαδικασιών διαχείρισης ε, μαζί με ε, την ανάγκη για αντικειμενική και αδέκαστη αντιμετώπιση των διοικητικών θεμάτων, την υπέρβαση προβλημάτων που προκύπτουν από συγκρούσεις ε, συμφερόντων κλπ. Και βεβαίως εδώ προκύπτουν και ζητήματα που αφορούν και την κοινοποίηση, τη διόρθωση κλπ. Ε, και τώρα μπορεί κανείς να βρει λύσεις ε, στα προβλήματα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι καλοπληρωμένους και καλά ενημερωμένους δικηγόρους που θα μελετήσουν ενδελεχώς όλα τα ε, θέματα και θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις. Ο γενικός κανονισμός που προτείνει το Κοινοβούλιο θα αφορά πράξεις βεβαίως θεσμών και οργάνων, αλλά θα αφορούν και τη διαδικασία λήψη απόφασης και άλλωστε η μελέτη επιβεβαιωτική δείχνει ότι ο κανονισμός αυτός ε, για τα διοικητικά θα μπορούσε να συμβάλλει ε, σε, ε, στη δημιουργία υψηλού επίπεδου προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς έτσι όπως είπε η συνθήκη της Λισαβόνας να πράξουν τα θεσμικά όργανα αλλά θα δώσει αυτήν την απαιτούμενη νομική βάση η Κομισιόν ε, Λισμονή να το αναφέρει αυτό. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η μελέτη αντικρύπου του Κοινοβουλίου δείχνει επίσης ε, ότι μια τέτοια πράξη διοικητικών ε, διαδικασιών θα μείωνε τον κατακαιρματισμό και θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ενοποίηση. Οποιαδήποτε διαδικασία απλούστευσης μπορεί να βοηθήσει την δημοκρατική εφαρμογή του νόμου και ε, ε, ε, την θετική εξέλιξη όσον αφορά τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον επόμενο ε, ομιλητή. Τον κύριο Ντύρκ Χούντιχ, Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ διαχείριση Κινδύνου. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να σα μιλήσω σήμερα εδώ και να λάβω μέρο ε, στην ακρόαση. Ήθελα να προσ προσαρτάγω στη, να προσφέρω στη συζήτηση κάποιες γενικές ιδέες από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διαχείρισης Κινδύνου. Ιδιαίτερως λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε ένα κυρίως θέμα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερο να έχει ή να μην έχει νομοθεσία για τις διοικητικές ε, διαδικασίες. Εγώ πιστεύω ότι για λόγους διοικητικούς, οικονομικούς αλλά και πολιτικούς πάνω απ' όλα είναι πολύ μεγαλύτερη αξία μιας, ε, νέας νομοθε... μιας νομοθεσίας διοικητικής παρά αυτό το οποίο μπορεί να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Καταρχάς το πώς βλέπει αυτή τη νομοθεσία ο κόσμος γενικότερα αλλά και οι επιχειρήσεις ευρύτερα τι θα σήμαινε με την νομοθεσία, σύντομα κάποιες ε, συστάσεις και το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Η διοικητική διαδικασία λοιπόν δεν είναι μια καινούρια ιδέα. Το 1767 ξεκίνησε η Σουηδία πρώτη χώρα ε, να ορίζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης στο Σύνταγμά της της εποχής εκείνης. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό ο νόμος για τις διοικητικές διαδικασίες, LAP. Γιατί, γιατί απλούστατα αποτελεί, ή μάλλον πρωταρχικά αποτελεί την ε, αυτόματη συνέχεια στα όσα έχει κάνει αυτή η τρέχουσα Επιτροπή Juncker ε, που σημαίνει ουσιαστικά ότι η δουλειά που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα έχει συνέχεια. Αυτό εξασφαλίζει κατά πρώτο λόγο ένα τέτοιο νομοθέτημα. Δεύτερον, ενισχύει ε, νομικό έρισμα, η νομοποίηση, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Τα ακούσατε ήδη νωρίτερα και από την προηγούμενη τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 46% των Ευρωπαίων πολιτών πολιτών δεν εμπιστεύονται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται βελτίωση και οπωσδήποτε η ε, νομοθεσία για τις διοικητικές διαδικασίες θα βοηθούσε να αντιμετωπιστεί γιατί θα θα ενισχύσει, θα, θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία. Τρίτον, βελτίωση διαχείριση κινδύνου και καινοτομία. Όπω ξέρετε, εγώ ε, ομιλώ πάντα υπό το πρίσμα τη διαχείριση κινδύνου ή της αντίληψης ε, της διακινδύνευσης. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, οικονομική δραστηριότητα, ανάπτυξη των βέλτιστων ε, προϋποθέσεων ώστε να ανθίσει η οικονομία, ώστε να μπορεί κανείς να προχωρήσει επενδύσεις. Και τι είναι αυτός ο όρος, η προϋπόθεση είναι η ασφάλεια δικαίου, κατά το οποίο οπωσδήποτε είναι απαραίτητο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, άλλωστε τον έφερε και η κυρία Χάουταλα. Πέραν λοιπόν της προοπτικής ε, που θα προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι εξυπηρετείται και ο στόχος της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας που έχει ορίσει ως ε, στόχο της η Επιτροπή Juncker. Ταυτόχρονα έχουμε το πεδίο και το φάσμα των δραστηριοτήτων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συν το χρόνο αναπτύξει και αναλάβει με αυτήν έστω την ε, κατακαιρματισμένη προσέγγιση, κατανοητό, αλλά αν κοιτάξουμε όλα τα καθήκοντα, άμυνα, έλεγχος συνόρων, ε, μεταναστευτικό, όλα αυτά τα θέματα τα οποία μπαίνουν μέσα στην ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, ε, αρμοδιότητες και πάλι ε, υπάρχει κίνδυνος αν κατά τρόπο κατακαιρματισμένο ρυθμιστούν. Θα μένουν κενά, θα διευρυνθούν υφιστάμενα κενά, θα καταστεί όλο και πιο ε, δύσκολο να γίνει η διαχείριση, να εξασφαλιστεί η διαχείριση αυτού του συστήματος καθώς θα είναι το όλο και πιο κατακαιρματισμένο. Και όσο οριμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται και πιο στεναρούς κανόνες για τον τρόπο λήψη των αποφάσεων και έκδοση των κανόνων. Άρα χρειάζεται λοιπόν ε, το, το εργαλείο εκείνο που θα επιτρέπει στα ευρωπαϊκά όργανα να διαχειριστούν το πιο περίπλοκο πεδίο και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και αυτό γιατί συζητούμε όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το πώς μπορούμε στο μέλλον να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Νέα ζητήματα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν ε, να ε, λειτουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτοί είναι οι τέσσερι βασικοί άξονε που δίνουν τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε την ε, διοικητική νομοθεσία. Το πεδίο επίση, Νωρίτερα αναφέρθηκε από τον κύριο καθηγητή ότι μπορεί να είναι λίγο πιο φιλόδοξη η δική μας η προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως στόχος θα είναι η κάλυψη των ε, εξουσιών αλλά και των ε, ε, εξουσιών προκύπτουν από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις 290-291 της συνθήκης, αλλά κάθε άλλη, άλλη πράξη, γιατί ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα δεν είναι ε, δεν είναι ζητήματα πρωτογενούς ε, δικαίου, αλλά δευτερογενούς που απορρέουν από κανονισμούς και πίσω από τους κανονισμούς και οδηγίες για την υλοποίησή τους, όπως το REACH που μπορεί να προκύπτει από ένα κανονισμό, αλλά έχει 1200 σελίδες κατευθυντηρίων γραμμών για την πρακτική υλοποίησή του, άρα χρειάζεται μια πιο συστημική προσέγγιση και όχι περιπτωσιολογική. Επίσης, η αξιολόγηση κινδύνου και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή πρέπει να ορίσουν αρχές πρότυπα για την ε, λειτουργία της διοίκησης, γνωστά, γνωστές αρχές στους πολίτες, ώστε ο πολίτης να αντιλαμβάνεται ποια δικαιώματα έχει. Έτσι λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε την ιδέα ενός ευρύτερου φάσματος από αυτά τα οποία συζητήσατε μέχρι τώρα σήμερα. Οφέλει και θα είμαι σύντομο. Ποιο θα ωφεληθεί. Πολύ σωστά είπε η συνήγορο του πολίτη ότι ο κύριο κερδισμένος από την υπόθεση αυτή είναι ο πολίτη και τελικά τι συνέπεια θα έχει αυτό, καλύτερες θέση εργασία, ποιότητα ζωή, ασφάλεια, ε, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, καλύτερη συμμετοχή του πολίτη στη διακυβέρνηση. Δεύτερον, και νομίζω ότι αυτό ήδη επισημάνθηκε, επίσης, τα ίδια τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. κερδίζουν καθώς ε, αντιμετωπίζουν ήδη κρίση αποδοχής και εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και εν τέλει, επιχειρήσεις και οικονομία. Η κυρία Χάουταλα ε, για μόνο μία φορά ε, φέρε το, τη λέξη ανταγωνισμό στην υπόθεση αυτή. Αλλά έχει τεράστια σημασία και δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο ένα περιθωριακό κομμάτι τη αξιολόγηση του τι θα προσφέρει αυτή η ασφάλεια για οποιονδήποτε, σαν περιβάλλον δηλαδή, για οποιονδήποτε θα ήθελε εδώ να επενδύσει. Εάν δεν υπάρξει αυτή η νομοθεσία, στην αντίθετη περίπτωση λοιπόν, διάβρωση, ε, σφαλμένες επιλογές, ε, επενδύσεις κακές και ούτω καθεξής. Τα ωφέλη νομίζω λοιπόν είναι σαφέστατα. Ξεπέρνουν δε κατά πολύ αυτά που ακούστηκαν νωρίτερα, γιατί τα 40 εκατομμύρια που ακούστηκαν είναι ψίχουλα δίπλα σε χαμένες ευκαιρίες, δίπλα σε προβλήματα και συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν, δίπλα στην ε, διατάραξη της λειτουργίας της κοινωνίας που μπορεί να προκύψουν. Όλα αυτά νομίζω ότι τα νούμερα αυτά, τα 40 εκατομμύρια, θα, μιλούσαν μόνο, θα ήταν νούμερα που αφορούν μόνο μία επιχείρηση. Μιλούμε για κάτι πολύ ευρύτερο σαν συνέπεια της απουσίας αυτής της νομοθεσίας. Ούτε καν μπορούμε να δούμε τις διαστάσεις του αυτή τη στιγμή και επιτρέψτε μου να περάσω στο γιατί έχουμε έρθει σήμερα εδώ. Καταρχάς η Επιτροπή έχει προβάλει αντιστάσεις στην ιδέα αυτή. Για τρεις λόγους κυρίως. κυρίως. Καταρχάς γιατί θεωρεί ότι αυτή η νομοθεσία θα οδηγήσει σε περισσότερες δικαστικές διαφορές. Αυτό το καλύψαμε. Δεύτερον θα περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια της διοικητικής, των διοικητικών αρχών. Τρίτον, γιατί μπορεί να προκύψει επιπλέον διοικητικό κόστο. Θα μου επιτρέψει τώρα να πω ότι είναι πολύ θεμητέ οι ανησυχίε αυτέ και επιφυλάξει. Θα τι απαντήσω όμω μία, μία προς μία. Ε, αύξηση των δικαστικών διαφορών. Αυτό νομίζω ήδη έχει καλυφθεί. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 100 χρόνια σε παιδοκρατών μελών έχει δοθεί απάντηση ξεκάθαρα και δεν υπάρχει κανένα λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προκύψει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει ε, αποδεδειγμένα από την ιστορία των ε, τουλάχιστον ε, τριών από τα 10, 6 ε, από τα 10 κράτη-μέλη. Ε, πλέον αυτό το επιχείρημα δεν είναι πιστικό. Μπορεί να το καταλαβαίνω γιατί προβάλλεται, αλλά δεν είναι πιστικό γιατί αυτό μα αποδεικνύουν τα κράτη-μέλη. Στερα από μια πρώτη περίοδο που θα χρειαστεί για την προσαρμογή, δεν υπάρχει αύξηση δικαστικών αγώνων. Δεύτερον, διακριτική ευχέρεια. Οπωσδήποτε η πρόταση αυτή δεν αποκλεί, δεν αφαιρεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποκλειστικό δικαίωμα στην νομοθετική πρωτοβουλία. Το να κρίνει κανεί ότι μπορεί να χάσει επίπεδο διακριτική ευχέρεια. Μπορεί να είναι κατανοητό μένα, αλλά όχι σοφό κατά με. Και θα εξηγήσω γιατί τι θα ήταν το... Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία. Θα είχαμε τις Βρυξέλλες εντό εισαγωγικών όπως την περιγράφουν οι ευρωσκεπτικιστές ε, που δεν θα ήταν υποχρεωμένε σε λογοδοσία, που θα ήταν ανεξέλεγκτε. Επομένω, με την νομοθεσία αυτή μπορεί η Επιτροπή να έχει και επιχειρήματα για να κάνει να σοπάσουν αυτέ οι φωνέ επίκριση. Άρα λοιπόν θα έχουμε όχι μία επιλογή που θα ακολουθούν απλώ ο ένα δημόσιο υπάλληλο μετά τον άλλον, αλλά μια επιλογή που θα γίνεται με βάση κανόνε, με βάση σαφεί διατάξει. Τρίτον, το επιχείρημα του κόστου. Το κάλυψα επίσης το κόστος του υφισταμένου συστήματος είναι πιστεύω πολύ υψηλότερο από αυτό που, που γνωρίζουμε, που μπορούμε να προβλέψουμε. Και οπωσδήποτε θα είναι θεαματικά τα αποτελέσματα της εισαγωγής νομοθεσίας. Και σχεδόν τελευταία παρατήρηση, συστάσεις της ε, υπηρεσίας μας. Έχουμε πολλέ, επομένω θα σας προτείνω να στρέψετε το βλέμμα στον τοπό μας, όπου είναι πολλές, όπου είναι καταγεγραμμένες όλες, αλλά εν συντομία τέσσερι μόνο συστάσει. Πρώτον, σαφές ε, διοικητικό ε, ευρωπαϊκό δίκαιο με νομοθετικά δεσμευτικέ προδιαγραφές. Δεύτερον, επίπεδο, ε, οπωσδήποτε επί, δυνατότητα, εξασφαλιζόμενη από το δίκαιο για ε, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων με την δυνατότητα ο πολίτης να διεκδικεί τα δικαιώματά του κατά τρόπο αποτελεσματικό. Τρίτον, δεσμευτικές προδιαγραφές και πρότυπα που να περιλαμβάνουν και τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις για τη δημόσια διαμοβούλευση, όπως είπε η κυρία O'Reilly. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ε, λιδία λίθο των, ε, του συστήματος του πώς υπηρετεί, σε τι βαθμό προσφέρει υπηρεσία αυτό το, αυτός ο διοικητικός μηχανισμός στον πολίτη και μέσα από τη διαδικασία αυτή των διαβουλεύσεων θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Τέταρτον, όλα τα σώματα και οι φορείς που έχουν ε, συμμετοχή θα πρέπει να εμπλέκονται και στην αναθεώρηση, τροποποίηση, ε, επανεξέταση της νομοθεσίας ε, όταν έρθει η ώρα για την αναθεώρησή της. Αυτά για το πεδίο που σας ανέφερα νωρίτερα, λέγοντας ότι είμαστε πιο φιλόδεξοι, όπω ακούστηκαν νωρίτερα. Τελευταία παρατήρηση, λοιπόν, γιατί είναι πολιτικά αναγκαία μια τέτοια νομοθεσία. Οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν διαρκείς πιέσει από τι ευρωσκεπτικιστικές φωνέ που οδήγησαν στον παραλογισμό του Brexit. Ένα τρόπο να ε, κάνουμε να σοπάσουν ε, οι φωνές αυτές που λένε ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν επαφή με, την, τον πολίτη, ότι η Επιτροπή είναι αδιαφανής, ε, δεν έχει λογοδοσία, είναι γραφειοκρατική, κλειστή, θα έβρισκαν απάντηση σε μια νομοθεσία για τις διοικητικές πρακτικές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν τεράστια ευκαιρία να δώσουμε αποτελεσματική απάντηση σε όλους αυτούς τους ευρωσκεπτικιστές, λέγοντας ακούσαμε τα επιχειρηματά σας και να η αποτελεσματική λύση. Έτσι λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε αυτές τις επικρίσεις και δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Εξού και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση και δεν πρέπει να παραμεληθεί. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ευχέρεια επιλογής, αλλά με καθήκον. Ευχαριστώ. Thank you, sir. As well, I'm sure that after... ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Λεναρντινή ε, θα μας τα πει ξεκάθαρα για αυτός όσον αφορά τη δική του οπτική γωνία από πλευράς ε, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς όπως αναφέρθηκε και στην εισήγηση από τον κύριο Αντιπρόεδρο εμείς ακούμε όλες τις απόψεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα της δημοσίας διαβούλευσης και τη αξιολόγησης των επιπτώσεων. Να σας αναφέρω τώρα κάποια ερωτήματα, κάποιες επιφυλάξεις. και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το ότι το διοικητικό δίκαιο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Βλέπουμε τα πράγματα αριαλιστικά. Άκουσα και τους σημερινούς ομιλητές και απεκόμισε την εντύπωση για το ότι ε, το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε ή όχι η νομοθεσία επί τούτο σήμερα έχουμε ένα πλέγμα ρηγητικών διατάξεων ανά τομέα και τώρα ερώτημα λοιπόν κατά πόσο όλα αυτά θα τα ενοποιήσουμε. Δεν με εντυπωσιάζει το πώς απήντησαν σε εκείνη την ε, έρευνα. Δεν συμμετάσχουν και τόσο πολύ. Τέλος πάντων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων όμως ε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και θα επανέλθω σε αυτό. Έχουμε μια σειρά ερωτημάτων και επιφυλάξεων όσον αφορά ε, το υλικό, όσον αφορά το βεληνικές αυτής της έρευνα και όσον αφορά την εκτίμηση για το, την περιπλοκότητα. Πρώτα-πρώτα θεωρούμε ότι είναι δύσκολο, αν όχι ρηψοκίνδυνο, σε ένα και μόνο νομοθέτημα να κάνουμε ένα συμπίλημα από στοιχεία διοικητικού δικαίου που αφορούν διαδικασίες ανακλάδου. Και άρχισε μια ματιά στο τι ισχύει στο κοινωτικό δίκαιο, ας πούμε τι ισχύει με οικονομικούς ε, ελέγχους όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη ή αν δείτε τι ισχύει με την νομοθεσία αντιτράστ, ε, τι εφαρμόζει δηλαδή η Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού, το δικαίωμα επιλογής της γλώσσας και το δικαίωμα σε απάντηση των πολιτών. Όλα αυτά ποικίλουν ως ρύθμιση ανάλογα με το σε τι τομέα αναφέρονται. Άρα υπάρχει ένα θέμα μεταξύ του οριζοντίου νομοθετήματος και της ιδιοτυπίες του κάθε τομέα. Τι θα πρέπει δηλαδή να παραμείνει το μεκαρνισμένο και τι και το κατευθυνόμενο. Ίσως θα πρέπει να μην τα πράγματα όπως ε, πρέπει. Γιατί η σημερινή ρυθμίση σχετίζεται με τις οδιοτυπίε του κάθε τομέα. Παράδειγμα, έχουμε την πρόταση του Κοινοβουλίου, όπου λέει για μια γενική πρόταση με 30 μερών για να ε, απαντήσει κανείς σε οτιδήποτε αίτημα. Και ισχύει το νομοθεσία ε, που προβλέπει συντομότερη προθεσμία για πρόσβαση σε έγγραφα είναι 15 μέρες της προθεσμίας. Τι θέλουμε, θέλουμε όλα να τα κάνουμε 30 μέρες, να τα εναρμονίσουμε και να ξέρουμε ότι και εν προκειμένου θα ισχύουν οι 15 μέρες. Μα μπορεί 30 μέρες για μια πλήρη έρευνα να είναι σύντομο όσον αφορά μια διαδικασία, παραβάση, κάποια τέλος πάντων καταγγελία σχετικά με κάποια παραβίαση. Και αν πάμε για ενιαία ρύθμιση τι σημαίνει αυτό, δεν θα υπάρχει εξαίρεση, μα τότε θα πρέπει να τροποποιήσουμε ε, τα πάντα και να έχουμε οριζόντια ρύθμιση σε επίπεδο διοικητικού δικαίου. Άρα όλα αυτά είναι συζητήσιμα και όλα αυτά είναι δύσκολο να ξεκαθαριστούν. Νομίζω ότι ο κύριος Τίμερμανς το είπε ε, δύο λίγων ότι υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά ακριβώς το τι είδους αποτέλεσμα θα υπάρχουν το, το νομοθέτημα τι θα είναι. Θα είναι κάποια ελάχιστα και θα μπορούν να υπάρχουν και εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις. Θέλουμε μια πλήρη εναρμόνιση, οπότε θα υπάρχουν ε, για το νομική νομοθεσία σημαντικές επιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά τα ένδικα μέσα, όλα θα μπουν σε αυτή την ενιαία ρύθμιση. Και κάποιοι μιλητές Οπότε θα πρέπει να είναι ευκολότερη η πρόσβαση στα θεσμικά όργανα αυτό όμως δεν είναι θέμα διοικητικού δικαίου. Είναι θέμα του να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για τα έγγραφα και τις διαδικασίες, να ανεβαίνουν όλα στο website. Κάπως διαφορετικό είναι αυτό το ζήτημα. Οπότε και εδώ υπάρχει προβληματάκι. Και κάποια από τα πράγματα που σας ανέφερα δεν είναι διοργανικά. Η κατεξιοδότηση πράξη για εφαρμογή αφορά τα κράτη-μέλη και όταν έχουμε την επιτροπολογία. Αλλά δεν μπορεί κάποιο άλλο να το κάνει αυτό. Και έχουμε κάποιου κανόνε για διαφάνεια, πρόσβαση έγγραφα, διαβούλευση, ε, για προκατακτική εκδοχή μέτρων. Όλα αυτά καλύπτονται από του κείμενου κανόνε. Άλλο θέμα είναι το πόσο περίπλοκο είναι το να γίνουν διαπραγματεύσει για κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε, διότι βλέπουμε ότι έχουμε προσπαθήσει κάποιες φορές να κάνουμε ε, εναρμόνιση της διοικητικής νομοθεσίας, οδηγούμαστε σε καθυστερήσεις, ας πούμε ο οργανισμός 1049 την πρόσθεση σε έγγραφα, προσπαθήσαμε να τον εξομοιώσουμε ή να τον εντάξουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας και να πούμε ότι ο οργανισμός αυτός θα ισχύει μόνο για Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μερικά άλλα θεσμικά όργανα τα οποία ειδικά κατονομάζονται. Αλλά τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα αυτό ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Και τώρα όμως έχει κολλήσει αυτή μας η πρόταση εδώ και πολλά χρόνια ε, στην νομοθετική διαδικασία. Ε, το 2016, άλλο παράδειγμα, είπαμε να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μητρό και έχει κολλήσει τις διαπραγματεύσεις. Οπότε βλέπετε ότι πρόκειται για συσύφη, για Τριτάνιο έργο τέλο πάντων. Πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να γίνουν. Γιατί προκύπτουν πάρα πολλέ δυσκολίε διοργανικά. Για να δούμε τώρα. Μια άλλη θετικότερη πλευρά, γιατί βλέπουμε ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων ανέδειξε μερικά ενδιαφέροντα σημεία και βλέπουμε πρώτα εδώ το θέμα των κανονιστικών υπηρεσιών που να εξομοιώνονται με τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι μια τάση που υπάρχει. Ε, υπάρχουν 30 τέτοιε κανονιστικέ ρυθμιστικέ υπηρεσίε, Μερικέ έχουν πολύ σημαντικέ αρμοδιότητε, αλλά το θεσμικό, η θεσμική αρχιτεκτονική αυτών των υπηρεσιών ε, προβλέπει να είναι ανεξάρτητες, να έχουν δική τους νομική προσωπικότητα, Κάποιες διατάξεις σε πρόσβαση στα έγγραφα δεν ισχύουν αυτές, μόνο αναλογικά εξαρτάται από τις υπηρεσίες, αν θα το εφαρμόσουν, οπότε βλέπουμε το ότι η αξιολόγηση είπε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Άλλα στοιχεία που ήταν ε, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα συγγνώμη, ήταν η ψηφιοποίηση, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο άσκησης της διοίκησης και του με τους πολίτες. Είπαμε ότι έχουμε τώρα ναι, μια καινούργια διαδικαϊκή πύλη. Μπορούν σε διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας οι πολίτες να συμβάλλουν και επίσης στο μέλλον. Θέλουμε αυτή η διάδραση να υπάρχει με κάποια μέσα άμεσης πρόσβασης του κόσμου. Άρα σε αυτό το σημείο συμφωνούμε με την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Okay. Thank you very much, Εγώ σας, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε περίπου 15-20 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως Πρώτα να ρωτήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν έχουν κάποια ερώτηση. Κύριε Αλιέφ, θέλετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακόμα πρέπει να πω ότι δεν βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την πρότασή μας για έγκριση ε, κανονισμού που θα θέσει κοινούς ε, κανόνες για την ε, διοίκηση. Ακούσαμε ότι έχει υπάρξει μια μελέτη και η μελέτη αυτή κατέδειξε ακριβώς τον κατακαιρματισμό ε, του, της διοικητικής νομοθεσίας. Ε, Μακρόσκελής διαδικασίες, μεγάλη επιβάρυνση, ε, φτωχή ελλειπή σε ποιότητα των απαντήσεων που παίρνουν οι πολίτες. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Στα πλαίσια του η ε, ιδιαίτερα περίπλοκου κανονισμού ε, του ισχύοντος όσον αφορά την ε, διοίκηση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαϊκός ο Ευρωπαίος Συνήγορος, καθώς επίσης και η ακαδημαϊκή κοινότητα δια, του εκπροσώ, δια των εκπροσώπων της έχουν καταδείξει μία σειρά διαδικασιών που πρέπει να εγκριθούν και να προχωρήσουν. Η λύση ε, ε, προέβλη, ε, προκύπτει καθαρά από την διαβούλευση που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο και από την μελέτη αντικτύπου. Ε, εδώ και δύο χρόνια λέμε ότι οπωσδήποτε με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι ελλείψεις στην νομοθεσία και θα κάνουν την νομοθεσία κατανοητή στο πνεύμα των πολιτών. Ταυτόχρονα θα δώσει διαδικασία ε, και αποδοτικότητα ε, του ευρωπαϊκού διοικητικού μηχανισμού. Μια ερώτηση στον καθηγητή Χόφμαν. Πιστεύετε ότι η πολιτική όθηση αυτή τη στιγμή ε, είναι κατάλληλη έτσι ώστε να προωθηθεί ε, αυτή η διοικητική πράξη. Ευχαριστώ κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό, κωδικοποίηση των διοικητικών διαδικαστιών, ε, πραγματικά ε, συγκλονιστικό το θέμα, κυρίως δε που εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαστε με αυτό, αλλά λίγο έχει προχωρήσει και εξελιχθεί. Έχουμε δύο στρατόπεδα τώρα, αυτοί που θέλουν την δημιουργία ενός τέτοιου κώδικα, νομίζω είναι η πλειοψηφία της Επιτροπής Νομικών ε, ε, Ζητημάτων, κυρίως δε ε, λόγω της θέσης και της επιμονής της κυρίας Χαουτάλα, καθώς επίσης αυτή θα είναι, είναι η θέση και της συνηγόρου κυρίας Χαουτάλα. Ε, απ' την άλλη πλευρά όμως, ε, και το διαπιστώνουμε για μία ακόμα φορά, υπάρχει και ένα άλλο στρατόπεδο. Εκεί που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας εξηγεί ότι η διαφοροποίηση, οι σε των υπηρεσιών είναι τέτοιου εύρους που ε, στην ουσία δεν θα καταφέρετε τίποτα και δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Άρα δεν θα προχωρήσουμε. Λυπούμε ειλικρινά γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με το θέμα αυτό κατηγορείται όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ε, ε, ένα διοικητικό τέρας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά φορά και εγώ ο ίδιος καταφεύγω σε αυτόν τον, ε, σε χαρακτηρισμό. Εν πάση περιπτώσει πρέπει πάντως όποια θέση και να έχει κανείς να αναγνωρίσει ότι είμαστε πολύ μακριά από τους διοικούμενούς μας. Θυμάμαι ότι είχε ακουστεί μία πρόταση πριν από πολλά χρόνια από τον κύριο Ούμπερ Λεγκάλ, ο οποίος ήταν ε, σύμβουλος ε, του γαλλικού κράτους και δούλευε για το Συμβούλιο, και σε μια άλλη δημόσια ακρόαση μας είχε ε, προτείνει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ανατμήματα, δηλαδή να μην κάνουμε ένα τόσο φιλόδοξο ε, κώδικα όπως ήταν η πρώτη προσπάθεια που κάναμε. Μας είχε ε, συμβουλεύσει να βγάλουμε τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον καθορισμό της διοικητικής πράξης και να ασχοληθούμε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως στην ίδια τη διοικητική πράξη πράξη περσέ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίε λοιπόν που έχουμε εμεί να πείσουμε την Κομισιόν, οι εμπειρογνώμονέ μα τι προτείνουν έτσι ώστε να μπορέσουμε παρόλα αυτά να προχωρήσουμε. Ε, thank ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και εγώ έχω ερωτήματα. Στον κύριο Λεραρντίνη. Αλλά να ρωτήσω το ένα από αυτά. Στην αρχή της παρεμβασίας σας, κύριε Λεαρντίνη, αναφερθήκατε σε δυσκολίες σχετικές ε, με δυσκολίες που σχετίζονται με τις 24 επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ε, σας κατάλαβα καλά. Ωραία. Α, κυρία Ντελβό, και εσείς θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν καθόλου να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, δεν θέλουν τίποτα να αλλάξει, αυτό είναι σαφές και προκύπτει σαφώς αντίθετα με τις απόψεις των βουλευτών του Κοινοβουλίου και των εμπειρογνώμων. Αλλά εάν κατάλαβα καλά αυτά που είπε η Κομισιόν, λέει ότι διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη δράσης όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις agencies. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε ε, αν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο για τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, τότε θα πρέπει να προκύψουν κάποιοι γενικοί κανόνες ε, πώς είναι δυνατόν να γίνει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση, να κάνουμε είτε κανονισμό είτε κατευθυντήρες γραμμές για τις agencies, αλλά να μην αγγίξουμε καθόλου ε, όλα τα υπόλοιπα στον ε, διηγητικό κανονισμό. Mm. Άλλη μία ερώτηση εγώ ήθελα να κάνω προς τον κύριο Χούντικ. Ε, ε, κύριε Χούντικ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Όχι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Εντάξει, όμως καλύτερα πρώτα να έχουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις των ε, βουλευτών και μετά να σας δώσω το λόγο. Παρατηρήστε κύριε Σχαουτάλα εκτός μικροφώνου. So you have been explicitly asked a question. Έχετε δηλαδή συγκεκριμένα δεύτερη ερώτηση. Ναι, βεβαίω το Κοινοβούλιο κάνει πολλέ προσπάθειες για να χτίσει αυτή την ε, ε, λογική και απόδειξη, αλλά υπάρχει το εξή που ανέφερε και ο κύριος Χοντήχη νωρίτερα. Υπάρχει η αποδουλία τη εμπιστοσύνη και τη αξιοπιστία, γιατί ε, υπάρχουν πολλές διαφορές από τη μία στην άλλη περίπτωση, κάτι που είναι περιττό, κάτι που οδηγεί τον πολίτη στο να μην καταλαβαίνει τι δικαιώματα έχει. Γι' αυτό είναι λάθος ο δρόμος αυτός για την Επιτροπή. Πρέπει η Επιτροπή να έχει και εκείνη μια διαδικασία, μια νομοθεσία διοικητικών πρακτικών σαν πρόταση, κατά το οποίο έχει κάνει μέχρι τώρα μόνο το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή δεν μιλήσει ακόμα για νομική βάση στη συνθήκη. Ο κανονισμό 41 του 1, 1049 του 1, ε, ορίζει κάποια στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα το ότι δεν αναφέρεται ότι προβλέπεται ρητά η ανάγκη για εγκαθίδρυση κανονισμού. Ο κανονισμός 1049 είναι παράδειγμα του πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προσπάθειές της, με τις προτάσεις της, ε, δεν κατάφερε τίποτε αρκετά ικανοποιητικό, γιατί προσπαθούσε να περιορίσει το γραφειοκρατικό φόρτο. Και το κοινοβούλιο δεν την ακολούθησε στον περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων. Επομένως, ε, ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα αυτός ο κανονισμός του τι θα έπρεπε να γίνει. Και συμφωνώ με την κυρία Ντελβό στο ότι όλο και περισσότερες ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, αποτελέσει και τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε εναρμονισμένους κανόνες. Τα τελευταία 15 χρόνια ε, έχουν θεσπιστεί υπηρεσίες αποκεντρωμένες που άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται σε διοικητικέ διαδικασίε, για τι οποίε θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει κοινό σύστημα κανόνων. Επίση, από τα όσα ακούω από την Επιτροπή, βλέπω ότι παρουσιάζει ψευδοδιλήμματα. Ε, μας λέει η Επιτροπή, αν δεν καταλαβαίνουμε αν πρέπει να υπάρξει σύγκληση ή εναρμόνιση. Εγώ θα έλεγα να κοιτάξει το κείμενο της πρότασης του Κοινοβουλίου η Επιτροπή του, της, πρό, της ε, πρότασης του 2016. Γιατί εκεί δεν αναφέρεται ούτε σε ε, κατελάχιστον, ούτε σε πλήρη εναρμόνιση, αλλά χρησιμοποιεί τον ε, κανόνα για την ε, κανόνα εναρμόνιση. Επομένω, εδώ έχουμε μία διάκριση, η οποία δεν σημαίνει ότι κάνω επιλογή μεταξύ γενικού ή ειδικού κανόνα. Μπορώ να έχω και τον γενικό κανόνα και τον ειδικό. Και εδώ η αναφορά στην ψηφιοποίηση και στα θέματα της ε, βελτίωσης της ε, νομοθετικής ε, διαδικασίας. Πάλι στο ίδιο επιχείρημα Το 2015 η Επιτροπή κατέθεσε 400 σελίδες ενδοτικού δικαίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας αυτής και με από τους ελάχιστους σε αυτή την υφήλιο που έχει διαβάσει τους κανόνες αυτούς προτινόμενους, όχι και όλες τις σελίδες βέβαια, αλλά εν πάση σε μεγάλο βαθμό. Ε, και βλέπω κάποια πρότυπα κανόνων ε, από τη θεωρία εδώ και χρόνια που οδηγούν προς, την προς το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή έναν κώδικα. Ε, το πρόγραμμα αυτό για το ενδοτικό δίκαιο νομίζω ότι θα μπορούσε λίγο πολύ να περιγραφεί σε 4, 5, 10 άρθρα απλά διατυπωμένα που θα αποτελούσαν τον μπούσουλα. Γιατί με την ε, ψηφιοποίηση των ε, διαγραμμικών θηρίδων, χωρίς να ενημερώνει όμως τον πολίτη, χωρίς να λέει γιατί γίνεται αυτή η απλοποίηση, αυτή η μετατροπή και ε, ε μήπως τελικά η μετατροπή έγινε γιατί κάτι λησμονήθηκε, γιατί ήταν εσκεμμένο και έπρεπε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Με το να μην εξηγεί λοιπόν στον πολίτη αφήνει ένα μεγάλο κενό και είναι σαφές. Ενώ με την κωδικοποίηση εξηγεί στον πολίτη ότι αυτή είναι η καταλληλότερη νομοθεσία και αυτό για να μην χάσουμε το μεγάλο δυναμικό που θα προσέφερε ε, ενιαίο διοικητικό νομοθέτημα. Γι' αυτό το λέω όχι ως πολιτικός αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής των ε, διοικητικών κανόνων και πάνω απ' όλα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα δικονομικά δικαιώματα των ε, πολιτών. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Έχουμε πολύ λίγη ώρα μπροστά μας. Στη θέση μας ακόμα. Παρακαλώ για ένα ή δύο λεπτά όποιος θέλει να ε, κάνει κάποια σχόλια. Ένα ή δύο λεπτά, ζητώντα συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρός με το χρόνο, αλλά έτσι δουλεύουμε εδώ. Η συνήγορος του πολίτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι με τη συζήτηση που γίνεται ε, και ως συμπέρασμα ε, ή ως σημείο εκκίνησης καλύτερα μπορούμε να δεχθούμε ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, επιθυμούν ένα καλό διοικητικό σύστημα. Ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει το διοικητικό δίκαιο αλλά να έχει πάντως μια γενική εικόνα για το τι σημαίνει δίκαιη μεταχείριση, η ταχεία εξυπηρέτηση και διεκπαιρέωση κτλ. Αν άκουει τη συζήτησή μας, οπωσδήποτε θα ε, αισθανόταν ότι τον έχουν πείσει τα επιχειρήματα των εμπειρογνωμών εδώ. Αλλά και του κυρίου Λεαρτίνη θα τον πείθανε. Ίσως πέραν από κάποια αμφιβολία για, το, ε, για τις διατυπώσεις ε, ότι α, υπάρχει πεδίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, κάποια σημεία λείπουν, υπάρχουν κενά κτλ. Δηλαδή μπορεί να τον μπέρδευε τον πολίτη η συζήτηση αν την παρακολουθούσε εδώ. Ταυτόχρονα όμως ρόλος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής είναι ακριβώς να διαλευκάνει αυτά τα σημεία ασάφειας και οπωσδήποτε θα ήταν κρίμα να μην δοθεί συνέχεια σε αυτή τη σημαντική συζήτηση και να καταλήγαμε σε ένα τέλμα ότως επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υψώνει φραγμούς στα όσα επιδιώκει το Κοινοβούλιο και οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπος επικοινωνία ε, συζήτησης μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής που ει βάθο να δίνει απάντηση στα μελήματα της Επιτροπής Αφενό ώστε και ο πολιτή όμω αφετέρου να μην ε, θεωρήσει ότι πρόκειται για μια ε, ιδεολογική αγκύλωση και ότι αυτή η εγκύλωση οδηγεί στο να μην ληφθούν οι αποφάσεις που πρέπει για να προχωρήσουμε σε ένα διοικητικό νομοθετικό σώμα που θα είναι προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χιούντιχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σοφά αυτά τα λόγια. Είμαι αναφανδόν υπέρ. Αν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει το status quo με κάθε τίμημα να διατηρηθεί. Αλλά για πόσο καιρό μπορεί να το κάνει, γιατί η συγκυρία δεν βοηθάει. Άρα θα πρέπει κάποιος ε, να, να είναι σε, σε ετοιμότητα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος. Θα πρέπει να ακολουθεί την τάση, τη ροή των γεγονότων. Τι γίνεται στις χώρες και δεν ανάγκη τα πράγματα να τα μπερδεύουμε τόσο πολύ αυτά τα άρθρα. Δεν, δεν είναι τόσο περίπλοκο το θέμα να είναι αδύνατο χειριστεί κανεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η βούληση για βελτίωση. Αυτό είναι η αφετηρία, η ιδέα για κάθε αλλαγή. Να δούμε δηλαδή τι πράγματα είναι δυνατόν να επιδέχονται έγκριση και κατόπιν να αρχίσει η προβληματική για το πώς θα το καταφέρουμε. Ε, αυτό μπορεί να είναι η κατάληξη τη σημερινή συνάντηση. Αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο για να ξεκινήσει αυτό το προτσές. Ένα ορόσημο. Σας ευχαριστώ σύντομα. Η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή μου καριέρα αφορά ακριβώς αυτό το θέμα. Για διάφορες χώρες, για διάφορα ε, συστήματα, ένομες τάξεις. Ε, ε, Βεβαίω και η ανταγωνιστικότητα και άλλοι οικονομικοί παράγοντες έχουν σχέση καθορίζουν την ποιότητα της διοίκησης περισσότερο από την ευκολία της επιχειρήσης, τη γραφειοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα. Ανοίξουμε μια ματιά τι γίνεται γύρω-γύρω. Έχω μαζέψει έγγραφα όλη μου τη σταδιοδρομία ανακοινώσεις, δηλώσεις, όσα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να υπάρχει ενιαίο νομοθέτημα, ενιαίος κώδικας ε, ε, για το διοικητικό δίκαιο. Αυτό έχει γίνει άλλο, γιατί με γίνει και εδώ. Βεβαίως και συμφωνώ ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα. Και ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα, το οποίο αποτελεί καμιά φορά φραγμό. Αλλά και τα κρατημέλη κάνουν πολλά. Τα είπε ο καθηγητής Χόφμαν. Τα περισσότερα κρατημέλη τα πέρασαν αυτά χωρίς να πάθουν και τίποτα. Χωρίς να υπάρξει κάποιο είδους αύξηση των ενδίκων διαφόρων. Τα είπε και η κυρία Ντελβό. Έχει μιλήσει για την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να αναγκαστούν οι Ιντερνετικές πλατφόρμες να διαχειρίζονται καλύτερα τη, τα παράπονα, τις καταγγελίες γιατί θα πρέπει να τσακώνεται με τα θεσμικά όργανα σχετικά με αυτά η κυρία Οράιλη. Μα έχουμε το Google, έχουμε ένα σωρό τρόπο τόσο ώστε κανείς υπεύθυνα να, να αντιδρά. Άλλο τώρα, όσον αφορά αυτό το θέμα με τις ε, υπηρεσίες και την εξομοίωση με αυτές, ε, σίγουρα αυτό το θέμα θα επανέρχεται, γιατί ακριβώς έχουμε κατάτμιση και όσον αφορά τις υπηρεσίες. Αλλά ισχύει αυτό το οποίο είπαμε τα, η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών στην διαμεσολαβήτρια αναφέρονται στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 60%. Άρα το πρόβλημα είναι δεδομένο. Δεν είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα είναι τελείως ξένη από αυτή την προβληματική και την ψηφιοποίηση. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχει κάποιο σημείο αναφορά σταθερά για να μπορεί τις διαδικασίες να τις ξεκαθαρίζει και αυτό να γίνεται παντού στην Ευρώπη για όλα τα θεσμικά όργανα. Α, και κάτι άλλο τελευταίο. Δεν προτείνουμε τίποτε ε, ακραίο. Είναι μινιμαλιστικές, συντηρητικές οι εναλλακτικές που προτείνουμε. Πιστεύουμε ότι αφού επιδέχεται το θέμα συμφωνία, μπορεί να βρεθούν και πιο τολμηρές λύσεις. Απλώς έχουμε περισσότερες αποδείξεις ότι μπορούν να αποδώσουν αυτές οι συντηρητικές λύσεις. Όχι στα ταμπού, όπως είπε ο κύριος Τίμερμανς. Άρα να κάνουμε βηματάκι προς τα μπρος και τότε θα δούμε ακτίδα ελπίδας για αυτές τις προτάσεις. Κυρία Εύα, Κυρία Εύα, συγγνώμη, έχετε κάτι να μας πείτε, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, θέλω να επανέλθω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Το είπαν και οι συνάδελφοι ότι χρειαζόμαστε ε, και ενωτομία. Δεν πρέπει να μείνουμε στην υπόθεση του status quo. Το πρόβλημα είναι δεδομένο, το είπε η διαβούλευση. Όλες αυτές τις λύσεις έχουμε. Και το είπαν και οι συνάδελφοι. η περιπλοκότητα. Δεν μπορεί να είναι λόγος του να επαναπαυθούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Και διάβασα τι είπαν οι πολίτες με αυτή την διαβούλευση. Θα πρέπει να κάνουμε τα προόδου, να βρούμε λύσεις, να μην κολλάμε ε, στις δυσκολίες, όπως το είπε ο συνάδελφος. Έχουμε νέα στοιχεία μπορεί τα κράτη-μέλη να έχουν πρωτοπόρο ρόλο. Να είναι παράδειγμα προς από πλευρά των ε, θεσμικών οργάνων. Αυτά τα κατέδειξε η διαβούλευση. Θα πρέπει να τα προσέξουμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα λεπτάκι, ναι, ναι, ναι. Επιβιώνω αυτά που είπε ο κ. Τίμερ μα ότι μα ενδιαφέρει να συνεχίσουμε αυτή την προβληματική. Νομίζω ότι πολλά μάθαμε σήμερα το απόγευμα και μα ενδιαφέρει η μελέτη των επιπτώσεων. Θα την μελετήσουμε οικονομική, πρακτική, νομική απόψεω όλα αυτά που ανέδειξε. Το θέμα παραμένει ε, εκρεμέ και θα μας απασχολήσει για άλλο. Τελευταία καταληκτική παρατήρηση, κυρία Χαουταλα, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς την υπηρεσία ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών ΣΥΠΙΑΣ. Βεβαίως και δεν ε, μπορείτε να έχετε όσο μεγάλο δείγμα χρειάζεστε τώρα που ζητήθηκε επισήμως να κάνουμε την έρευνα για την αλλαγή της ώρας το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ε, θα πάρουν πολύ μεγαλύτερο δείγμα τώρα. Είναι κάτι άχρηστο. Ε, σε αυτή την έρευνα θα έχουμε εκατομμύρια απαντήσεων. Παρόλα αυτά. Ή ισχύουν αυτά που είπε η συνήγορο στον πολίτη. Ότι είναι αυτές οι βασικές αρχές που πρέπει να διεύουν τη διοίκηση. Χωρίς αυτές τις αρχές ο πολίτης δεν ξέρει τι γίνεται. Ευχαριστώ την Εμίλη ότι ήρθε η ώρα να τα συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεργαστούμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Τόσες απαντήσεις δόθηκαν σήμερα το απόγευμα πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να προλιάνουμε το έδαφος για την επόμενη επιτροπή. Και η Φινλανδία κατά σύμπτωση δεύτερο εξάμεινο του 19 θα ασκεί την Προεδρία. Και σας υπενθυμίζω συνεχώς ότι εμείς ήμασταν οι εμπνευστές το 1998. Γι' αυτό και έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και είδατε όλα αυτά που λέξανε για το 18ο αιώνα και τη διοίκηση ε, στην Σουηδία, αφορά και εμάς, γιατί τότε ανήκαμε στην ε, Σουηδία, ήμασταν με τη Σουηδία. Και μετά είχαμε και το 766 τότε που δόθηκε μια όθηση στην ανταγωνιστική οικονομία των χωρών εκείνων. Όχι 18ο 8 8ο αιώνα. Ευχαριστούμε καθηγητά που μας είπατε για την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη στενή σχέση ε, που έχουν με σταθερότητα των θεσμών. Άρα, το κυδετικό δίκαιο είναι συνεκτική ουσία, ούτω ώστε όλα αυτά να συντεριάζουν. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και σωστά τα είπε ο κύριος μας που ευτυχώς ήρθε να μας μιλήσει. Αρχίζουμε αρχίσουμε τη συνεργασία για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προτελέσουμε το έδαφο για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα λέει ο πρόεδρο. Σα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές, τους εμπειρογνώμου που ήταν σήμερα μαζί μας, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Ουραϊλή και βεβαίω και τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Τίμερμαντ, ε, για τι αρχικέ του παρατηρήσει. Ε, ε, νομίζω ότι πραγματικά κάναμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα βήμα επιπλέον προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Dear colleagues, we continue by item 29. Uh, Περνάμε στο επόμενο θέμα μας και καλώς την κυρία Ελισπέτα Μπιένκοφσκα, Επίτροπο της ε, Ιστορικής Αγοράς Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βιομηχανίας. Σας είχαμε καλέσει πριν από μερικού μήνε ε, στο πλαίσιο βέβαια του διαρθρωμένου διαλόγου. Με χαρά σας βλέπουμε σήμερα εδώ. Στις 29 Νοεμβρίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση μέτρων ε, για την ε, τεχνολογία της πληροφορίας με διάφορες ανακοινώσεις για τέτοια θέματα καθώς και κατευθύνες γραμμές για την οδηγία IPRED, για την επιβολή των δικαιωμάτων Τη ε, πνευματική ιδιοκτησία Μέχρι τώρα δεν είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, Επομένω, είναι καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και τα θέματα αυτά. Και εντωμεταξύ 28 Μαου υιοθέτησε μια πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, επικουρική για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα ε, τον οποίο επίσης έχει την αρμοδιότητα η Επιτροπή μας, οπότε μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας στο θέμα αυτό. Θα πρότεινα λοιπόν να πάρετε το λόγο εσείς για 15 λεπτά. Να ακούσουμε μετά τους συναδέλφους της Επιτροπής μας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά τους και εάν το επιτρέψει ο χρόνος και το ενδιαφέρον μπορούμε να κάνουμε δύο γύρους ερωτήσεων και απαντήσεων. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ιδιαίτερα ε, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα ενημερώσω για την ε, δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πραγματική ιδιοκτησία και βέβαια θα ήθελα να ενημερώσω και για άλλα θέματα που θα σας ενδιαφέρουν ασφαλώς. ξεκινώ αναφερόμενοι σε δύο στοιχεία. Καταρχάς, τομείς ένταση της Πνευματική ιδιοκτησία που είναι 56-3 εκατομμύρια σε επίπεδο ΑΕΠ. Δύο από τι πέντε θέσει εργασία είναι θέσει εργασία σχετικέ με την ε, πνευματική ιδιοκτησία. 90% των εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έχουμε είτε μεμονωμένου τίτλου για το εμπορικό σήμα και σχέδιο και σε ένα βαθμό το δίπλωμα ευρεσιτεχνία και κανόνε για το απόρριτο και κανόνες που καλύπτουν το SPC και άλλα θέματα που θα σας διευκρινίσω αργότερα, καθώς και κανόνες για την επιβολή των ε, δικαιωμάτων ε, πνευματική διοκτησία. Πρόσφατα έγινε η ολοκλήρωση, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση του εμπορικού σήματος. Πριν από ένα μήνα περίπου τέθησε ισχύ στα κράτη-μέλη η οδηγία για το επαγγελματικό απόρριτο. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι ορίζει πρότυπα, αλλά δεν, δεν επαναπαυόμαστε. Ξεκινούμε με νέες πρωτοβουλίες, μια πρωτοβουλία παραδείγματι για τη στρατηγική ε, πνευματικής διοκτησίας για τα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, πακέτο ε, μέτρων με την επιβολή αλλά και τις, τις άδειε ε, τα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνία πάλι στο πλαίσιο τη πνευματική διοκτησία και πρόταση για την εξαίρεση SPC. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο θεματολόγιο για την επιβολή των δικαιωμάτων. 2,5% είναι το παγκόσμιο εμπόριο ε, των προϊόντων απομίμησης ή πειρατικού χαρακτήρα. 5% ε, όλων των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αξία 85 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα προϊόντα απομίμησης που κυκλοφορούν στις αγορές μας. Βεβαίως μια νομοθετική προσέγγιση θα ήταν πολύ χρονοβόρα και δύσκολο να επιβληθεί. Είχαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία με μηχανισμούς ε, διεκδίκηση αποζημίωση σε περίπτωση παραβιάσεως των δικαιωμάτων αυτών. Στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούν, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ως ε, σημείο μέτρησης ή μέτρο στάθμισης ε, αυτές τις ε, κατευθυντηρίες γραμμές. Ελπίζουμε φυσικά να μας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πνευματικής Διοκτησίας, Βιομηχανικής Διοκτησίας με την ε, ε, εμείς με τη συνεργασία μας σε διαφορούς παραγόντες από τη βιομηχανία, δικαιούχους κτλ. Έχουμε επίσης μια διαδικασία αυτορύθμισης σε σχέση με την ε, διαδικτυακή διαφήμιση που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους διαφήμιση αν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας και λοιπά δικαιώματα σε όρους εμπορικής και έτσι ελπίζουμε ότι η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ε, θα αποκοπεί από ένα από τα κύρια έσοδά της. Ε, το Νοέμβριο του 2017 καταθέσαμε αυτή την πρόταση ε, για την πνευματική διοκτησία, σύνολο προτάσεων καλύτερα, που ορίζει και πρότυπα ουσιας, θεμελιωδών βασικών διπλωμάτων. Και έτσι έχουμε και τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, για τις ε, ε, μικρές επιχειρήσεις κτλ. Έτσι λοιπόν... Μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πολύ καλή αντίληψη του τι σημαίνει ε, δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση και διαπραγματεύσεις ε, περιπτωσιολογικά. Καλούμε τους εμπλεκόμενους φορούς, φορείς να προσέλθουν στις συνομιλίες ε, με τρόπο θετικό. Βεβαίως θα δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και σαφήνεια θέλουμε να προσφέρουμε για την ανάπτυξη του ίντερνετ των πραγμάτων, της, 5G, της τεχνολογίας 5G, των αυτόνομων ε, χημάτων, Θεμάτων δηλαδή πολύ σημαντικών για το εγγύς Σε συνέχεια, στις ε, μέχρι τώρα πρωτοβουλίες, θεσπίζουμε τώρα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που στόχο θα έχει να βελτιώσει την αξιολόγηση και την αδειοδότηση αυτού του τύπου των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και θα πούμε θα οριστεί από αυτή την ομάδα ποιες, ε, ποια είναι τα διπλώματα που έχουν αυτές τις βασικές ε, προδιαγραφές για να μπορούν σε ε, όρους θεμητούς να χρησιμοποιούν ε, την τεχνολογία που κρύβεται πίσω αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας οι επιχειρήσεις μας. Για τα έσπισης, λοιπόν, σας έχουμε πει ότι ε, υπήρχε η πρόταση αυτή για να υπάρξει παρέκκληση SPC. Την καταθέσαμε 28 Μαΐου. Πρόκειται για μια παρέκκληση που αφορά μόνο τις εξαγωγές και θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει ε, ε, προϊόντα γενετικής ε, παραγωγής, γενικής παραγωγής και βιοϊσοδύναμα να έχουν ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και ευκαιρίες για είσοδο σε τρίτες ε, αγορές. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουν πολύ καλύτερο σημείο κίνησης στη διαδρομή τους ε, στις αγορές αυτές τα προϊόντα μας. Ταυτόχρονα αυτό θα βοηθήσει και τις επενδύσεις. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας Βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερο είναι το μερίδιο της αγοράς για τα βιοεισοδύναμα και τα γενετικά προϊόντα. 80% αναμένεται να είναι όγκος τους το, 20%, το 2020 και 85% σε παγκόσμιες πωλήσει. Ωστόσο δεν περιμένουμε τώρα ε, στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ε, γενικής παραγωγής και βιοεισοδύναμα να ανταγωνιστούν μέσα στις διεθνείς αγορές. Είναι πολλά τα ιατρικά προϊόντα των οποίων θα λήξουν από το 2020 και μετά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Έτσι λοιπόν ανοίγει μια αγορά 95 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κόσμο ολόκληρο. Και άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξή ερώτημα. Ποιο ωφελείται από τις νέες ευκαιρίες ε, που θα προσφέρουν οι αγορές Εμεί θέλουμε αυτά τα φάρμακα, ε, τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, τα δικά μας, ε, να είναι ε, μεταξύ των πρωτοπόρων για να μην αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο της απώλειας των εγκαταστάσεων παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας, της ιατροφαρμακευτικής βιομηχανίας συνολικά, των θέσεων εργασίας. Ακούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή στις διαβουλεύσεις όλους τους εμπλεκομένους, τις ανησυχίες, τις προσδοκίες τους. Βάσει αυτών που ακούσαμε προτείναμε μια ισορροπημένη, σταθμισμένη και αναλογική πρόταση για την ε, παρέκκληση έσπιση. Χωρίς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αλλάζουμε τη διάρκεια της προστασίας της βιομηχανικής ε, ιδιοκτησίας για τα φαρμακευτικά το, χωρίς να αλλάζουμε το όλο σύστημα SPC, διατηρώντας γενικά την, το σύστημα της ευρεσιτεχνίας και των SPC, ε, που άλλωστε προάγουμε σε όλες μας τις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις, χωρίς καμία πρόθεση να το αποδυναμώσουμε. Η προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής διοκτησίας στην Ευρώπη είναι πολύ ισχυρή και ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την πρόταση αυτή, η οποία εξασφαλίζει στο πλαίσιο της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων τη δυνατότητα για παραγωγή των προϊόντων αυτών στην ε, ευρωπαϊκή αγορά, μόνο εάν πρόκειται αυτά να εξαχθούν, εάν είναι δηλαδή οι γενικής παραγωγής ή βιοεισοδύναμα, και πρόκειται να εξαχθούν σε χώρες ε, στις οποίες επιτρέπεται η πώλησή τους, εκτός όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε. Εδώ λοιπόν μπορούμε να διασφαλίσουμε και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξασφαλίσουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίω σε εξαγωγέ για τον βιομηχανικό μας κλάδο. Οφελούμε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη θα δουν ωφέλη. Επιβεβαιώνουμε την θέση της Ευρώπης ως άξονα για τα φαρμακευτικά προϊόντα και την φαρμακοβιομηχανία αλλά θέλω πως λίτως να κατασοφές ότι δεν έχει καθόλου στόχο αυτή η νομοθεσία να ε, προτιμήσει ή να ευνοήσει ένα κλάδο της ε, ε, βιομηχανικής παραγωγής. Γι' αυτό και έχουμε ορίσει πολύ αυστηρές προδιαγραφές και δεσφαλιστικές δικλείδες, όπως είναι η κοινοποίηση, όπως είναι η προσήκουσα επιμέλεια και άλλα, με αποτέλεσμα το διαφάνεια στην αγορά για το ποιος παραγητή και για τους στόχους. Έτσι αποφεύγεται και ο κίνδυνος. Να παραστρατήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που θα έπρεπε να την χάνουν προστασία τη πραγματικής ε, διανοητικής ιδιοκτησίας. Ελπίζουμε ότι προς όφελος όλων των πλευρών και παραγόντων του κλάδου θα μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα αυτή η απόφαση. Στήριζομαι στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας ειδικότερα και το θέμα αυτό νομίζω πολύ σύντομα συζητήθηκε σε μια πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο εχθές ή προχτές και έμαθα ότι υπήρξε γενικά έκφραση υποστήριξης από όλες τις χώρες της Ευρώπης για την πρόταση αυτή. Ελπίζουμε ότι και η Αυστριακή Προεδρία θα προωθήσει γρήγορα την πρόταση. Και θα ήθελα να πω και δύο λόγια, κλείνοντας, για το εργαλείο πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς. που πιστεύω μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή σας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα φόρου αποφυγή, σε θέματα ε, ετοιμάτων για ενημέρωση που έχουμε ε, μετατρέψει σε εργαλεία για την πολιτική και ως Επιτροπή, εγώ ως Επίτροπος, είδαμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι δυνατότητες, όπως σε παραδείγματι με τα σκαρδαλά για τους με το ντίζελ, τα διαδικά προϊόντα και άλλες ε, προτάσεις, είδαμε ότι πρέπει να έχουμε στη θέση μας αξιόπιστα δεδομένα. Όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Είχαμε κατευθυντήριες γραμμές και ασφαλιστικές δικλίδες για την ε, προστασία και την ακρίβεια των δεδομένων με προσεκτική ανάλυση νομικής βάσης οπωσδήποτε. Η νομική βάση από την ενιαία αγορά 114 της συνθήκης είναι ένα σωστό εργαλείο, αλλά υπογραμμίζω ότι αυτό προτάθηκε ως εργαλείο γιατί η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν όλοι τηρούν τους ίδιους κανόνες. Η επιλογή του 114 ήταν μια σαφής και για μας την Επιτροπή αλλά και για την νομική μας υπηρεσία και ξεκάθαρη επιλογή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στη συζήτηση αυτή. Χρειαζόμαστε την συμμετοχή του. Εξασφαλίζει άρρωστα το 114 και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις νομοθετικές διαδικασίες. Η Επιτροπή όμως Εταιρική αγοράς από ό,τι αντιλαμβάνομαι προτείνει μια διαφορετική νομική βάση που θα απέκλει το Κοινοβούλιο από την όλη συζήτηση, πράγμα το οποίο μου φαίνεται και λάθος και παράλογο. Ο εισηγητής της Επιτροπής ΕΜΚΟ μου το ανέφερε αυτό και με πάση ειλικρίνεια σας το μεταφέρω ως το δυνατόν πιο κομψά. Αλλά οπωσδήποτε χωρίς το Κοινοβούλιο και σε ένα θέμα τέτοιο, όπως αυτό της ιστορική αγοράς, δεν είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε αλλιώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπη για αυτά που μας είπατε και έχουμε τώρα την δυνατότητα να, δώσουμε, να υποβάλουμε ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Dank. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα να διατυπώσω δύο ερωτήσει για τα SPC. Ίσως, βέβαια, με τις, ε, άμα πούμε σε βαθμό λεπτομέρεια, ε, μπορεί να δείτε ότι είναι δύο-τρει. Τελικά, όχι μόνο δύο. Έχω πάντω την αίσθηση και η νομική υπηρεσία άλλωστε το διεπίστωσε. Ε, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι με την αλλαγή του συστήματος ε, συρρυκνούνται τα δικαιώματα και βλέπουμε ότι προκύπτει ένας κίνδυνος απαλωτρίωσης χωρίς αποζημίωση. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές ε, ε, λεπτομέρειες. Ή να με πείσετε με περισσότερες λεπτομέρειες ότι δεν βλέπετε κίνδυνο για απαλωτρίωση χωρίς αποζημίωση. Δεύτερον, τι θα εννοούσατε εσείς, τι θα βλέπατε ως κόκκινη γραμμή σε όλη αυτή τη ε, διοικητική διαδικασία και συμπληρωματικά. Στα θέματα συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου πιστεύετε ότι σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Κυρία Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν περιορίζουμε τα υφιστάμενα δικαιώματα ε, η εξαίρεση θα αφορά μόνο τα SPC τα οποία δεν έχουν ακόμα αποδοθεί. Ε, βεβαίως υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ε, ωστόσο, οπωσδήποτε ευθυγραμμίζονται με όλες τις συμφωνίες, τις υφιστάμενες δηλαδή συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αυτά. Ε, α, ναι, και εδώ μου λέει η μου ε, οι ή μελλοντικέ συμφωνίες ελεύθερου ε, εμπορίου, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να αντιτίθεται στις ισχύουσε ή μελλοντικέ ε, free trade agreements, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Κύριε Φως. Για τι κόκκινε στο πλαίσιο της νομοθεσίας, πού θα βλέπατε κάποιες κόκκινες γραμμές εσείς. Μπορούσε να προχωρήσει κάτι τέτοιο σύντομα, να κλείσει μέσα στην τρέχουσα θητεία. Και μια και τον Απρίλιο μάλλον δεν θα είμαστε πλέον εδώ, ίσως τον Μάρτιο-Φεβρουάριο να πρέπει να κλείσει. ή τουλάχιστον αυτό να στοχεύουμε σε σχέση με το κομμάτι που θα αφορά την ε, απόφαση του Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε η Επιτροπή να δώσει κάποιε ενδείξει για το ε, ποιε θα ήταν οι δικέ τη κόκκινε γραμμέ για την νομοθετική διαδικασία. Απάντηση. Πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω συγκεκριμένε κόκκινε γραμμέ. Πάντω αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα αυτό και μετά από τη συζήτηση στο Συμβούλιο είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση ότι δεν υπάρχουν δηλαδή σημαντικά έτσι σημεία σύγκρουσης. Μονάχα ένα κράτος μέλος είχε κάποιο προβληματισμό για να σας αποκαλύψω και κάτι όσον αφορά τις προτάσεις αυτές. Αυτό που προσπαθούμε ακριβώς και αντιμετωπίζοντας ε, τις ανησυχίες όλων των πλευρών και για τα γενικά και για τα biosimilars και τα ε, ε, καινοτόμα στοιχεία. Πιστεύω ότι εμείς κάναμε μία πολύ ισορροπημένη πρόταση. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχουν κάποια σημεία σύγκρουσης. Επίσης η οικονομική βάση και η ανάλυση του συνόλου ε, είναι πολύ καλά, δεν έγινε στο πόδι. Ε, και πραγματικά μας πήρε μήνες μέχρι να κάνουμε την πρόταση αυτή το timing, ε, η χρονική στιγμή ε, και ο ρυθμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για μας και δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα με τούτη την πρόταση. Τώρα, τι να σας πω, η ισορροπία, ναι, θα μπορούσε να είναι κόκκινη γραμμή. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κόκκινη γραμμή. Δηλαδή να μην ε, ε, γύρουμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι κόκκινη γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Ζήφκα. Θα ήθελα να πω το εξή. Προφανώς ε, κόκκινη γραμμή θα μπορούσε να είναι τα οικονομικά ζητήματα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τα οικονομικά ζητήματα δεν είναι τα μόνα που έχουν σημασία. Σημαντικό είναι και το θέμα της ασφάλειας, να διασφαλίσουμε δηλαδή την ασφάλεια. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία έχουν ίδιο βάρος και σημασία εάν τροποποιήσουμε ε, την, ε, ε, την νομοθεσία μας για τα SPCs, ε, τότε ε, ίσως θα πρέπει να έχουμε και κάποια προτίμηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δρούν εντός της επικρατείας του, του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια κόκκινη γραμμή όλα, οτιδήποτε, οτιδήποτε βελτιώνει την κατάσταση των επιχειρήσεων στις ε, τρίτες χώρες, γιατί μπορεί να προκύψει μια τέτοια ε, θέση εάν ε, δεν δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν, αυτό θα μπορούσε να είναι με μια κόκκινη γραμμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπεραμεινθούμε της φαρμακευτικής μας αγοράς. Ξέρουμε ότι οι γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά Μπορεί να φοβηθούν, ναι, αλλά με την ίδια ευκολία μπορούν να πάρουν ε, μία, ε, μία άλλη ε, οδό διαφυγής που είναι το να βγάλουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ε, εργοστάσια τους. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές που δεν μπορούν να σταθούν ως ίσον προς, ίσως με τους ε, ε, γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας. Κοιτάξτε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε αμέσως μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές, ε, εάν βεβαίως ε, και το Συμβούλιο έχει τη διάθεση, αλλά από ό,τι μας αποκάλυψε και η κυρία Επίτροπος, φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα αγγλικά εάν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Θέλω να είμαι πολύ σαφής οι δικέ μα προτάσει, ε, τι αποκαλώ τι προτάσει μα ισορροπημένε, γιατί λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία τη κατάσταση. Βεβαίω δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου ο ανταγωνισμό, ε, καθώ επίση και καινοτόμε ε, φαρμακευτικέ βιομηχανίε μέτρα την Ευρώπη να εξαφανιστούν. Αυτό είναι φυσικά μεγάλη μα προτεραιότητα. πιστεύω ότι η πρότασή μα είναι καλά ισορροπημένη, καλά στοχευμένη ε, ναι, είναι γεγονός ότι μπορεί αυτοί που ε, είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουν κάποια ε, αυξημένη, κάποιο αυξημένο ανταγωνισμό από τους εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, κυρίως όσον αφορά τα biosimilars και όσον αφορά και τα γαλλικά φάρμακα, τα γενώσιμα και αυτά. Αλλά Πιστεύουμε ότι η κατάσταση, η θέση έτσι όπως την παρουσιάζουμε είναι θετική, είναι win-win. Και επομένως δεν ε, έχουν τρομερά προβλήματά ούτε οι originators ούτε τα biosimilars. Ε, πιστεύω ότι ε, εδώ μιλάμε και για ένα δις για τις εταιρείες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, θέσεις εργασίας για υψηλά εξειδικευμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Φως, θέλετε και άλλη ερώτηση. Ich wollte nur noch mal nachfassen. Ναι, προσπαθώ όμως να καταλάβω σε σχέση με αυτό το κίνδυνο της επαλωτρίωσης ε, έχει η Επιτροπή αναλογιστεί εάν υπάρχει αυτός ο νομικός κίνδυνος ή όχι. we think that this risk just Πιστεύουμε ότι αυτό περιλαμβάνεται στην πρότασή μας. Δεν, δεν, προ... Συγγνώμη, δεν περιλαμβάνεται αυτό στην πρότασή μα. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ε, ε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να χάσουμε, να χαθεί αυτή η προστασία. If Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, να σας ε, ευχαριστήσουμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε και συζητήσαμε αυτά τα τόσο σημαντικά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Βιενκόφσκα. Εγώ είχα προετοιμαστεί για πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Πάντως, σκεφτείτε την πρόταση. Εντάξει, εδώ έχει κλείσει, αλλά θα είναι κρίμα να μην έχουμε το κοινοβούλιο στο πλευρό μας γι' αυτό. Thank you. Thank you so we are finishing? No, not yet. Not yet, not yet. No. Thank you very much.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 Okay, dear colleagues, we may continue. Ο Πρόεδρος, να συνεχίσουμε συνάδελφοι. Γιατί διακόπτει. We can continue by item. Συνεχίζουμε, Λαβάνη. Πρόεδρος, έχουμε τώρα το θέμα υπαριθμών 27 εξέταση της εκθέσεως για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιές του ενωσιακού δικαίου. Η συγκίτρια είναι η κυρία Ροζιέρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και να σας επαναλάβω ότι αισθάνομαι ικανοποίηση που έχουμε αυτή την νομοθετική πρόταση τώρα που το συζητήσουμε. Είναι αυτό το ζήτημα των καταγγελόντων Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που άρχισε το θέμα να ανακοινείται και έχουμε πρόοδο στο θέμα και βέβαια στο μέτωπο της φοροδιαφυγής αλλά και για τους ε, καταγγελόντες οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτή τη διαδρομή ξεκίνησε πέρσι με μια έκθεση και θέλουμε τώρα να υπάρξει νομοθεσία σχετικά με αυτά τα πρόσωπα. Η πρόταση Επιτροπής είναι πολύ ενθαρρυντική και έχουμε αυτό το σχέδιο κειμένο που σας παρουσιάζω και θα επιστώσετε εδώ, προτείνω κάποιες τροποποίησεις στο αρχικό κείμενο, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις καταγγελίες χωρίς να φεύγω από το πνεύμα του κειμένου, δηλαδή την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και την αναγνώριση του ρόλου αυτών των προσώπων. Επίσης, να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην ε, πληροφορία και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Έχουμε διάφορα στοιχεία στο κείμενο. Πρώτα-πρώτα το πεδίο εφαρμογή. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα. Άρα χρειάζεται όσο γίνεται ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή. Και γι' αυτό και ξανατονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση της Επιτροπής που προβλέπει ευρύ και οριζόντιο πεδίο εφαρμογή. Άρα μένουμε σε αυτό το πνεύμα. Πάντως έχουμε κάποια επιφύλαξη ακόμα. Έχει ήδη αναδειχθεί το θέμα το ότι δεν περιορίζεται στις παράνομες πράξεις αλλά στις πράξεις τις παράνομες δηλαδή αλλά σε οτιδήποτε, ε, σε οτιδήποτε πράξη παραβλάπτει το δημόσιο συμφέρον όπως και στο Lux Leaks οι σχετικέ καταγγελίε δεν ήταν με τη στενή έννοια παρανομές πράξεις, αλλά ε, εστρέφονται κατά του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Άρα χρειάζεται νομοθεσία σχετική. Επομένως να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή, να λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλυφθούν επομένω και οι σχετικές καταγγελίες. Τώρα όσον αφορά τους καταγγέλλοντες να εξασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται από το κείμενο. Ε, μπορεί να έχουν κάποια πληροφορία που να καλύπτεται από τη σχετική οδηγία και θα μπορούσαν να είναι στόχοι για αντίπεινα. Άρα παράσχουμε εγγύησεις προστασίας. Και για τον καταγγέλλοντα και για όποιους τον βοηθούν. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Α, ή βεβαίως και οι ασκούντες ερευνητική δημοσιογραφία. Και αυτοί θα πρέπει να καλυφθούν γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών δολοφονιών δημοσιογράφων τελευταία. Άλλο σημαντικό θέμα που θέλω να κάνω μια αλλαγή είναι κάτι για την καταγγελία. Με απασχολεί το ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το στόχο της οδηγίας να προστατεύσει επομένω τους καταγγέλλοντες. Άρα την ώρα της καταγγελίας θα πρέπει να ξεκινάει η προστασία. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, να έχουμε κάποιο στεγανό μηχανισμό, ξεκάθαρο, που να προσαρμόζεται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Όπως και να γίνεται η καταγγελία λοιπόν. Μέσα στην υπηρεσία απ' έξω κλπ. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα χρονικά πλαίσια της κάλυψης ε, της καταγγελίας και να είναι τόσο άμεση η αντίδρασή μας τόσο ώστε να προλαβαίνουν οι ε, καταγγελόμενοι να ξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης να προβλέπεται η παροχή συμβουλών ε, και μέσα στην υπηρεσία τους αυτών που θέλουν να προβούν σε καταγγελίες. Η λογική της προστασίας τους επιβάλλει εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους. να μην ε, προκτούνται συνθήκε που να οδηγούν σε τροχοπέδι και σε αποφυγή της καταγγελίας. Έτσι το ειδούμε σε περισσότερες καταγγελίες. Η αποτελεσματικότητα της ε, καταγγελίας ε, είναι ένα θέμα εδώ. Στο κείμενο της Κομισιόν. Έχει ιεραρχήσει τα θέματα εδώ η Επιτροπή, ούτω ώστε κάποιο θέλει να καταγγείλει. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να το πει στον εργοδότη μέσα στην υπηρεσία του και κατόπιν μπορούμε να πάμε μέχρι τρει μήνε όσον αφορά την επεξεργασία τη καταγγελία. Και αν δεν ικανοποιηθεί, μπορεί τότε να πάει ε, εξωτερικά. Πάμε στους έξι μήνες τότε και αν πάλι δεν γίνει τίποτα, μπορεί να ε, το δημοσιοποιήσει αυτό που θέλει να καταγγείλει. Έτσι όμως παραβλάπτεται η ουσία της καταγγελίας. Έτσι είναι πιο εύκολο να υπάρξουν αντίπεινα. Και έτσι είναι πιο εύκολο να καταστραφούν στοιχεία. Θα πρέπει να έχουμε πρώτα-πρώτα στο μυαλό μας ως προτεραιότητα την προστασία του καταγγέλλοντα και της καταγγελίας. και να μην είναι δική του ευθύνη η τήρηση αυτής της ιεραρχικής κατα ε, τέλος πάντων υποβολής της καταγγελίας. Άλλωστε υπάρχει εδώ ανισότητα μεταξύ του ενός οργανισμού, μιας υπηρεσίας και από την άλλη μεριά ενός φυσικού προσώπου που έχει το θάρρος να ρισκάρει ε, το να παραμεθεί στη δικαιοσύνη ή να υποστεί κάποιο είδους ε, αντίπεινα. Αν δεν κάνουμε αυτά που σας λέω τότε χάνετε το νόημα της ε, προστασίας. Άρα θα πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτές τις επιμέρους ε, σκέψεις να δούμε πιο πολλές εναλλακτικέ. να υπάρχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τις διάβλους, ε, τους διάβλους της καταγγελίας. κίνητρα, οπισθοβουλία, δεύτερη σκέψη που λέγαμε όσον αφορά τον καταγγέλλοντα και αυτά θα πρέπει να καλυφθούν για να μην αντιβαίνουν στο σκοπό ε, της ε, νομοθεσίας αυτής για την προστασία δηλαδή. Περιεχόμενο τώρα της προστασίας πέραν των διάβλων της καταγγελίας. Πώς θα τον προστατεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Η ε, γενική απαγόρευση αντιπίνων, σωστά τα πρόταση της Κομισιόν. Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό αυτών που σκέφτονται να προβούν σε αντίπεινα. Έχουν πολλές ιδέες, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε εδώ κάποια αποκλειστική απαρίθμηση για το τι μπορεί να γίνει ε, και άρα θα πρέπει να είναι ενδεικτική απαρίθμηση το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα αντίπεινα. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης, λέει η Κομισιόν, όσον αφορά τα αντίπεινα. Αυτό προστατεύει, αυτό λαμβάνει υπόψη το συσχετισμό των δυνάμεων. Αυτό θα πρέπει να το εγκρίνουμε. Τώρα το θέμα της ανώνυμης καταγγελίας. για το θέμα αυτό θα πρέπει να έχουμε πρακτική προσέγγιση. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και αντιστοιχούν στο ότι ο καταγγέλων πολλές φορές είναι πολύ ευάλωτος για να κάνει επώνυμη καταγγελία. Αλλά το θέμα δεν είναι τώρα πώς θα ρυθμίσουμε, πώς θα οργανώσουμε τέτοιες καταγγελίες. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν κάποιος κανιονών καταγγελεί και κατόπιν αποκαλύπτει την ταυτότητά του ενώ θέλει να παραμείνει ε, ανώνυμος, να μην στερείται του περιθωρίου, το να μην στερείται της δυνατότητας της προστασίας. Άλλο αδύνατο σημείο είναι η του. Υπάρχει η επαγγελματική του σχέση, ε, υπάρχουν τα αντίπεινα, υπάρχει η παραπομπή του στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως το ότι υπάρχει και το θέμα της απομόνωσης αυτού του καταγγέλλοντος. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να έχουν βέβαια την ευελιξία στη ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάθε είδους ε, πλαισίωση, συμβουλής του καταγγέλλοντος. Βέβαια να προσέχουμε να μην φτάσουμε σε αβάσιμες καταγγελίες. Και αναλόγα με τις συνθήκες να ακολουθεί το πιο σωστό διεύλο καταγγελίας ο καταγγελών. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, υπάρχει ο ρόλος των ΜΚΟ, τα συνδικάτα, γίνονται των πολιτών, πολλοί μηχανισμοί. Όλα αυτά θέμητα. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τον ρόλο αυτών των καταγγελόντων και να μπορεί να υπάρχει επιλογή του διάβλου της καταγγελίας ε, ανάλογα με την κατάσταση. Είπαμε θέματα οικονομικά, είναι θέματα ε, νομικά, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή η απομόνωση, η αίσθηση του ότι κανείς είναι μόνος έναντι κάποιου ισχυρότατου οργανισμού. Και αυτό δυσκολεύει την ε, πράξη της καταγγελίας. Είναι ψυχολογικό το φράγμα αυτό. Χρειάζεται επίσης ασφαλεία δικαίου. Δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει την καταγγελία και γι' αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε επιπλέον κυρώσεις σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας. Μα ήδη προβλέπονται κυρώσεις. Η συκοφαντία διώκεται. Επιπλέον ποινικέ κυρώσεις δεν βοηθάνε για την προστασία των καταγγελαντών. Έτσι κι αλλιώς είναι στριμωγμένοι. Είπαμε να ε, ισορροπήσουμε τα πράγματα. Άρα εάμα κάνουμε πιο αυστηρές τις κυρώσεις, αυτό έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για το να γίνει η καταγγελία. Άρα σε αυτό το σημείο να απαλληφθεί το κείμενο. Αυτό είναι η πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης ε, αφού γίνει η αξιολόγηση των επιπτώσεων του κειμένου, αφού αξιολογηθούν τα κενά του νομοθετήματος και να δούμε και συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις που εντωμεταξύ θα ανακύψουν. Αυτά προτείνω. Ε, τώρα όσον το χρονοδιάγραμμα, οι συνάδελφοι καταθέσουν τις τροπολογίες τους μετά τις θερινές διακοπές 6 6-9 το μεσημέρι είναι η προθεσμία. Πιέζει λίγο το χρονοδιάγραμμα αλλά στη Γιούρη πρέπει να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο και έχουμε και τον τρίμερη διάλογο που μπορεί εκεί να συζητηθεί ε, το συντομότερο η πρότασή μας. Αυτά και περιμένουν υπόμονα, συνάδελφοι, τις προτάσεις Thank you very much. Ευχαριστώ. 6 Σεπτεμβρίου προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Συνεδρία των σκιωδών προηγείται. Και θα είναι στα θέση σε όλες οι μεταφράσεις μέχρι τότε. Κύριος Γκυρό. Ναι, Πρόεδρε. Έχει πέρασει και η ώρα, έχουμε και πολλά θέματα ακόμα μπροστά μας. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για άλλη μια φορά ευχαριστώ τη Βυργινία, όπως άλλωστε πάντα κάνω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. 100% συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις της και επί της ουσίας και ως προς την φιλοσοφική θεώρηση αλλά και ως προς την νομική τοποθέτηση. Περιμένω να ακούσω τι έχουν να πούν και οι άλλες ομάδες. Εν τω μεταξύ όμως θέλω να διαβεβαιώσω τη Βυργινία για την υποστήριξή μας. Κάποιες τροπολογίες θα υπάρξουν αλλά υποστηρίζουμε πλήρως τις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να αποχωρήσω. Πριν φύγω σας εύχομαι πολύ καλές διακοπές. Τελευταία η συνάντησή μας αυτή πριν από τις θερινές διακοπές. Ξεκουραστείτε καλά και να σας ξαναβρω, να ξαναβρεθούμε όλοι. ξεκουραστεί και φρέσκοι το Σεπτέμβριο. Παραδίδω το θρόνο στην κυρία Τελβό. Okay, I immediately give the floor to και δίνω το λόγο στην κυρία Γιούντελαντ αμέσω. Καλώς ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Βιργινία για την πρόταση αυτή. Είναι πολύ σημαντική δουλειά, καλή δουλειά, θα φέρει σημαντικές αλλαγές για την Ευρώπη. Και είναι απαραίτητο βεβαίως να σημειώσουμε το όφελος που θα έχει για τους πολίτες. Είναι απαραίτητο η κοινωνική εταίρη, το ότι καλύπτονται οι κοινωνικοί εταίροι στο άρθρο 4.1. Αλλά βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε τους τρεις διευκρινήσεις, συγκεκριμένα δηλαδή ε, μνήα των σωματείων των συνδικαλιστικών, και γενικά την προστασία του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, στην παροχή νομικής υποστήριξη όποιον αποφασίζει να καταγγείλει κάτι του οποίου έλαβε γνώση από την υπηρεσία του και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιούτε. Ποιο θες πολύ σύντομα. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και περιμένω τις επόμενες συζητήσεις μετά τις διακοπές. Σημείο 31, ανταλλαγή απόψεων. Α, 30. Ψηφιακά εργαλεία και διαδικασία στο εταιρικό δίκαιο. Έχουμε και τον εισηγητή εδώ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Θα τον ε, παρακαλέσω λοιπόν, αν δεν έχει αντίρρηση, να λάβει πρώτο το λόγο. Ναι, ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες ψηφιακές στο εταιρικό δίκαιο. Ε, το 31 είναι αυτό όμως. Mm make maybe an uh, your your yes and this και σας ευχαριστώ για την υπομονή. Thank you very much, Mrs. President. Uh, If I... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχετε ε, κόψει ας πούμε το το θέμα σε δύο ε, το, ε, και το πρώτο είναι οι συγχωνεύσεις κλπ. Ε, και μετά το δεύτερο κομμάτι είναι τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς το είχαμε δει από κοινού. Ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Εγώ έχω μια ημερήσια διάταξη με δύο στοιχεία. Από την Έχω ένα θέμα Digital Tools και ένα θέμα Cross-Border Conversions και Mergers. Θέλετε να τα, ε, αλλά τα συζητούμε μαζί, μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί. Αυτό είναι πολύ καλό, λέει ο κύριος Δημητριάδης, γιατί ε, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς δουλεύουμε ε, για το θέμα από κοινού. ζητώ όχι εγώ ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, αλίμονο. Ε, έρχομαι από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή ε, και δουλεύουμε λοιπόν ε, για αυτά τα δύο εργαλεία, ευελπιστώντας ότι θα ολοκληρώσουμε την μελέτη των εγγράφων αυτών τον Οκτώβριο. Εγώ προσωπικά προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και εκπροσωπώ τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η νομοθετική δέσμη ε, θα ξεκινήσω με τα ψηφιακά εργαλεία, γιατί είναι πολύ σημαντικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, ε, αντιμετωπίζονται σαν ένας πολύ περίεργος κόσμος εδώ στις Βρυξέλλες. Πρέπει να σας πω ότι όταν εμείς στην Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για πραγματικά μικρές και μεσαίες. Δεν χρησιμοποιούμε τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί βάσει του ορισμού αυτού ε, καλύπτονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ε, ε, αλλά έχουμε 19-20 ε, εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι ακριβώς μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Σε γενικές γραμμές να σας πω ότι θετικά διακύμεθα απέναντι σε αυτή την δέσμη και χαιρόμαστε και πραγματικά ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας έδωσε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά ζητήματα, τα ψηφιακά εργαλεία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κόστος γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις πραγματικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολύ συχνά ως εκπρόσωποι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουμε τις δυνατότητες, δεν έχουμε και τις δεξιότητες που χρειάζονται, δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να μην πω όπλα, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε στην ψηφιακή, ψηφιοποιημένη κοινωνία. Κατανοείτε καλά ε, εύκολα γιατί αν ε, είμαστε σε ένα μικρό μαγαζί, σε μια μικρή επιχείρηση, σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτούς τους ιδιοκτήτες που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο προσπαθώντας να ε, κρατήσουν ε, ε, την εταιρεία τους μέσα σε ένα τόσο αντίξο περιβάλλον. Πραγματικά αυτοί πολλά έχουν να κερδίσουν εάν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι πολύ σημαντικά το ε, το θέμα αυτό θα μπορέσει να μειώσει την γραφειοκρατία και θα δώσει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταγραφούν εύκολα ε, χωρίς ε, αυτούς τους σημαντικούς περιορισμούς που έχουμε τώρα. Από την άλλη πλευρά μας ενδιαφέρει πολύ να χρησιμοποιηθούν σωστά ε, και με ασφαλή τρόπο αυτά τα ψηφιακά εργαλεία από τις επιχειρήσεις. Ε, περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς ε, η καταχώρηση των επιχειρήσεων και τα ψηφιακά εργαλεία θα είναι στην πραγματικότητα, στην πράξη. Όσον αφορά τώρα τις διαστηνοριακές μεταστροφές, να σας πω ότι είναι λίγες και αναφέρομαι εδώ για, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, πολύ λίγες είναι αυτές οι οποίες έχουν το θάρρος ε, να περάσουν τα σύνορα, να διαβούν αυτόν τον Ρουβίκονα έτσι ώστε να κάνουν ε, δουλειές εκτός των συνόρων τους. Επομένως για πρώτη φορά αυτή η νομοθεσία είναι πολύ σημαντική. Για πρώτη φορά παίρνουμε ένα σημαντικό θετικό βήμα το οποίο εμείς υποστηρίζουμε γιατί ιδιαιτέρως θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την ενιαία αγορά, θα δοθεί πλέον η δυνατότητα στις πραγματικά μικρές επιχειρήσεις να δουλέψουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός συνόρων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη. Έχουμε δύο εισηγητέ. Γιατί είπαμε ότι εμείς για οργανωτικούς λόγους ε, ξεχωρίσαμε τα δύο θέματα. Ο κύριος Ζήφκα πρώτος. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία για την χρήση των εργαλείων που πλέον έχουν καταστεί απαραίτητα στην ψηφιακή μας οικονομία. Ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία να συστήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πρόταση η οποία ιδιαίτερα απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξασφαλίζει τη δυνατότητα της καταχώρησης εταιρεία. μέσω του διαδικτύου με ταχύρυθμες διαδικασίες μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Είναι μια πρόταση που περιμένανε και η αγορά και οι επιχειρήσεις και όλες οι έρευνες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα μέσον το οποίο ήταν απαραίτητο να προκύψει με τις ε, σχετικές αναθεωρήσεις της νομοθεσίας. Αυτό περιμένουν οι επιχειρηματίες μας. Επίσης η πρόταση Επιτροπής ε, ορίζει και κάποιες προϋποθέσεις που θα ήθελα να αναφέρω. Προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει δεκτή η κατάθεση της ε, αίτησης καταχώρησης στο διαδικτύο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν τα συστήματα ταυτοποίησης για να γίνουν σεβαστές διαδικασίες online. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν σαφή ε, στοιχεία ταυτοποίησης. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να ε, καταχωριστεί ή να καταχωρήσει εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζει ποιε είναι οι προποθέσει, ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσει για να γίνει ε, σεβαστή η διαδικασία. Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αμφισβήτηση. Τρίτον, πάλι υποχρεωτικό στοιχείο, θα πρέπει να είναι αυτό της μίας και μοναδικής αίτησης καταχώρησης. Από έναν ιδιώτη μπορεί να κατατεθεί μόνο μία αίτηση για την καταχώρηση μίας μόνο εταιρεία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χρειαστεί να ε, υποβάλει διαφορετικές αιτήσει, διαφορετικές αρχές του κράτους μέλους ο ενδιαφερόμενος. Μία μόνο κατάθεση αίτησης. Επίσης, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ε, παραμέτρους ενιαίες για την ε, διαγραμμική κατάθεση, ένα ενιαίο πρότυπο ή μοντέλο του, της αιτήσεως και σαφείς αρχές και κανόνες για την ε, ταχεία και διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών. Πάνω απ' όλα αυτό δεν πρέπει ε, ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των αρχών και των επιχειρήσεων, τη επιχείρηση που ενδιαφέρεται να καταχωριστεί. Εννοείται ότι αυτό δεν πρέπει να προξενήσει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, γιατί έχουμε να κάνουμε πολύ μικρέ επιχειρήσει, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε να κάνουμε με τη ραχοκοκαλιά τη εσωτερική αγορά, τη ενιαία αγορά. Επίση, πρέπει να εξετάσουμε και ενδεχόμενε απειλέ που μπορεί να υποκρύπτονται μέσα σε αυτόν τον τρόπο καταχώρηση, κάποιου κινδύνου ενδεχομένω και να τους αντιμετωπίσουμε, να τους προλάβουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η κατάθεση της αίτηση για την καταχώρηση μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, εάν, εάν εγείρει βάσιμες υποψίες η αίτηση αυτή, εάν φαίνεται ότι δεν είναι τελείως καθαρή η καταχώρηση. τότε μπορεί να ε, επιτρέψει μία επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και μάλιστα ε, ενώπιος ονοπίο. Μετά υπάρχει και η λύση των ενοποιημένων μητρών, δηλαδή μπορούν τα κράτη να επαληθεύουν εάν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας υπάρχει περίπτωση να έχει καταγραφεί σε, κάποιο, σε κάποια μαύρη λίστα άλλου κράτους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σχέδιο της οδηγίας ως προς την ε, καταχώρηση των ε, επιχειρήσεων δεν κάνει παρέμβαση σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, μόνο και καταχώρηση μιλούμε εδώ ε, και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα κράτη-μέλη σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλους. Ορίζεται. Βεβαίως το κράτος μπορεί να έχει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και μπορεί και να απαιτήσει την παρέμβαση συμβολογραφικής αρχή. όσο συνήθως γίνεται μάλιστα στα κράτη. Επομένω, αυτή η δυνατότητα για την ε, ε, παρέμβαση συμβολογράφου στη δικασία καταχώρηση, δεν ε, χάνεται, δεν αποκλείεται. Από την πρόταση της Επιτροπής, λοιπόν, εγώ καταλήγω ότι είναι μια καλή πρόταση, είναι απαραίτητη οπωσδήποτε. έχοντας παρακολουθήσει και τις ε, διαβουλεύσεις επίπεδο επιτροπής, ε, βλέπω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε επίπεδο νομοθετικό, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να καταχωρίζονται με τη διαδικασία αυτή. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι τηρούνται όλες τις προδιαγραφές ε, που μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια ε, της ε, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή αναγνώρισης ταυτότητας όπως και του ελέγχου των ελέγχων σε περίπτωση κάποιας παράβασης της νομοθεσίας. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στις διατάξεις της οδηγίας. Ε, Κλείνοντα, θα ήθελα να πεθύνω έκκληση να ξεκινούν το χειρότερο δυνατό οι εργασίε για το θέμα αυτό, ώστε να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία στη διάρκεια ακόμα τη δική μα θητεία. 3 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, έχουμε την κατάθεση της πρότασης, έκθεσης. 10 Σεπτεμβρίου την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών παρουσίαση της έκθεσης πρώτα, μετά κατάθεση προλογιών και ενδεχομένως μετά ε, την ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε το θέμα των, ε, με το θέμα των μετατροπών σχολάσεων και διαιρέσεων. Εξαιρετικό είναι το θέμα. Εγώ ήθελα να ακούσω όλους τους χειώδεις για να δω ε, τι θα <clears throat> καινούριο στοιχείο θα ανέφεραν όσον αφορά το θέμα αυτό. Ναι, εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ε, ε δύο διαφορετικές ε, δύο διαφορετικά θέματα, συγγνώμη. Και νομίζω ότι εδώ καλύπτονται κάποιες παρόμοιες ανάγκες ε, για να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε το θέμα γρήγορα αλλά αποτελεσματικά. Γρήγορα γιατί πρέπει να ε, προχωρήσουμε με τα παραδοτέα. Η Επιτροπή μας ε, έχει ε, πολύ καιρό ασχοληθεί με το θέμα ε, και είναι σημαντικό με αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν τώρα. Και νομίζω ότι το ίδιο μπορώ να πω και εγώ με αυτό που είπατε τελειώνοντας την παρέμβασή σας και στις συγχωνεύσεις, σε μετατροπές ε, ε, και εξαγορές. Ε, το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε κι εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο να ε, υποβληθεί ε, και από τη δική μας πλευρά η πρόταση. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και input από την κοινωνία των πολιτών, να ξέρουμε ποια είναι και η δική τους άποψη. Όσον αφορά την ίδια την, ε, το ίδιο το θέμα, είναι σημαντικό που έχουμε την πρόταση και είναι σημαντικό να έχουμε νομική ε, βεβαιότητα, γιατί μόνο με νομική, νομική βεβαιότητα ε, μπορούμε να βοηθήσουμε και να προστατέψουμε τους εμπλεκόμενους. Τώρα, τα θέματα τα οποία ε, θέλω να βάλω στο τραπέζι είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τις ε, ε, ρυθμίσεις, τις τεχνητές ρυθμίσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου η, ο, ε, νόμος που διέπει, η νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις είναι τόσο περίπλοκος, είναι τόσο περίπλοκη νομοθεσία, είναι ένα πλαίσιο τόσο περίπλοκο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μην ε, επιτρέψουμε περιθώρια για καινούριε τεχνητές ε, ρυθμίσεις ε, που στην ουσία μπορεί να αποτελέσουν ε, πρόσκομα στην ελεύθερη μετακίνηση. Τώρα το ερώτημα είναι είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα της ε, ε, επιχείρησης. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι θετική η απάντηση. Την ε, καθαρή, ε, την καθαρή δραστηριότητα της επιχείρησης θα πρέπει να δούμε. Γιατί αυτό αποτελεί επίκεντρο ένα άλλο θέμα το οποίο θα θέλαμε να αναφέρουμε σε σχέση με την έκθεση είναι όλα αυτά που σχετίζονται με τη διαδικασία. Ε, βλέπουμε τι προτείνει η Κομισιόν, ε, εστιάζεται στην διαδικασία. Δεν θα μπορούσαμε όταν ασχολούμαστε ε, με αυτές τις συγχωνεύσεις και λοιπά, δεν μπορούμε να βασιστούμε στη γενική οικονομική δραστηριότητα και μετά να γίνει λίγο λιγότερο περίπλοκη η όλη διαδικασία, να την κάνουμε λίγο λιγότερο ε, περίπλοκη. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα ε, διευκολυνθεί η διαδικασία και αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το ρόλο των, ε, του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητος όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις εθνικές αρχές οι οποίες αντιμετωπίζουν το θέμα. Χρειαζόμαστε πραγματικά αυτόν τον εμπειρογνώμονα. για το σκέφτομαι. Αυτό που δεν θέλω είναι να ανοίξω μια νέα διαδικασία ή ένα νέο πεδίο ε, για ε, τις ε, επιχειρήσεις ή ένα είδος φόρουμ όπου θα ε, γίνεται συζήτηση. Όταν υπάρχουν εθνικές αρχές που έχουν τις σωστές αρμοδιότητες, ναι, οπωσδήποτε μπορεί να έχουν αυτές έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ρωτάω τους υπόλοιπους συναδέλφους και τέλος, δεν διστάζω να πω ότι είναι σημαντικό να μην προσπαθήσουμε ε, να ε, περιορίσουμε τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν ήδη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα, δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα, αλλά αυτά είναι τα ε, στιγμή επί των οποίων θα εστιάσουμε εμείς την προσπάθειά μας και την θέση μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εύελιν, κυρία Σταράς θέλει το λόγο και τον έχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Λουίστικ Γκράντες που είναι ο σκιώδης εισηγητής για την ε, οδηγία αυτή. Και μου είπε να σας πω ότι χρειάζεται η τροποποίηση της σχετικής νομοθείας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε επίσης στις ε, προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, κοινωνικές, οικονομικές, επίσης να βοηθήσουμε στην κινητικότητα όλων των επιχειρήσεων να βοηθήσουμε το εμπόριο. Βεβαίως και το θέμα είναι περίπλοκο γιατί υπάρχουν ε, νομοθετικές δυσκολίες και διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Και τα σημαντικά θέματα δεν είναι προστασία των εργαζομένων, ακριβώς όπως είπε η συνάδελφος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και θα πρέπει επίσης οι πιστωτές ε, αλλά και οι μέτοχοι να μην θυγούν από αυτήν την ε, δομική, διορθωτική αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να προσταθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες και θα πρέπει να έχουμε τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς, τους πιο απλούς και έτσι θα έχουμε εξοικονόμηση δαπανών για όλες τις επιχειρήσεις. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι το ότι χρειάζεται να είναι σταθερό το νομοθετικό περιβάλλον τόσο ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη προς την ε, ενιαία αγορά. Και ακριβώς αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση της ε, απάτης. Είναι σημαντικό, λέει, να μπορέσουμε να έχουμε έναν ορισμό του τι πάει να πει τεχνητή συμφωνία και να μην έχουμε αναδιάρθρωση κάποιας εταιρείες που να γίνεται κακόπιστα, να γίνεται επιλεκτικά και να έχει σκοπό τη φοροδιαφυγή. Οπότε έτσι να καταπονεμήσουμε και να μειώσουμε τον ε, αριθμό των εικονικών εταιρειών. Θα πρέπει να έχουμε επίσης ε, για να προχωρήσουμε στη σύνταξη του οριστικού κειμένου και κάποια γνωμοδότηση από κάποιους ειδικού. Δεν είναι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ αναγκαίο αυτό το μέτρο. Συγγνώμη, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Αλλά είναι αναγκαίο το μέτρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και ευχαριστώ και τον προσκεκλημένο μας από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Πολύ χρήσιμο το να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας κύριε. Όσον αφορά τώρα τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία σε σχέση με το τερικό δίκαιο, ο σε εισηγήτρια. Αλλά να σας πω τι, τι λέω για αυτές τις δύο συμφωνίες. Νομίζω αυτό είναι μια δέσμη μέτρων που πρέπει να την επεξεργαστούμε εδώ. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες για το εταιρικό δίκαιο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξυγχρονίσουμε το δίκαιο αυτό. Με την ψηφιοποίηση αυτή θα μπορέσουν να καταχωρούνται σε μητρό ιντερνετικά οι εταιρείε. Είναι σημαντικό να χτενιστεί αυτή η οδηγία όπως πρέπει, να αντιμετωπίσουμε απάτη, ε, τις εικονικές εταιρείε και ε, αυτού του είδους η καταχώρηση των εταιρείων είναι αξιόπιστη. Τα συνδικάτα ήδη έχουν ε, διατυπώσει κάποιε επιφυλάξεις σε σχέση με το να γίνονται όλα ιντερνετικά και ε, όχι μόνο από φυσικά πρόσωπα, από νομικά, αλλά και από φυσικά γιατί έχει δείξει πρακτική πόσο περίπλοκο είναι να αποδειχθεί το ότι μια λαδαπή εταιρεία έχει ιδρυθεί με σύνομο τρόπο. Γιατί είχαμε τόσα σκάνδαλα, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks. Η εμπειρία κατέδειξε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανειληφθεί ποιο είναι ο ιδρυτή τη εταιρεία, ποια είναι η ταυτότητά του, όταν δεν υπάρχει νομικός ε, ή νομοθετικός έλεγχος. Και όταν ιδρύεται κάποια εταιρεία μόνο για ε, λόγους φοροδιαφυγής και άλλα επιλήψεμα. Τι λέει ο συγκριτής ε, της ΟΚΕ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας από αυτού. Επίσης, φυσικά και θέλω να ακούσω και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες, τις συγχωνεύσεις, τις ε, διαιρέσεις. Συμφωνώ με την Εμίλη Ρίγνερ. Αυτή η πρόταση για τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για να τα εξετάσει είναι κάτι το νέο, νέα ιδέα για πολλά εθνικά συστήματα. Έτσι υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με την χώρα ε, αφετηρίας έτσι έχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαιοποίηση, θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές ρήτρες εξασφάλισης. Να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές διεκδικήσεις. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις ΜΜΕ και αυτά να τα δει ο εμπειρογνώμονας. Αν δεν θέλουμε παράκαμψη του νόμου, να μην εξαιρέσουμε κανέναν από αυτόν τον έλεγχο. Γιατί το θέλει αυτό η Κομισιόν. σε Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις. Δύο λεπτά έχουμε ακόμα, λέει ο πρόεδρος. Μετά θα σταματήσει η Γερμηνία αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Μήπως θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Mrs. Chair. My name is Maya. Law Unit in... Από την Γενική Διεθνήση για τη Δικαιοσύνη σας ομιλώ. Και το μόνο ζήτημα που προκύπτει είναι εάν ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να δικαιούται να χρησιμοποιήσει το ε, ηλεκτρονικό εργαλείο καταχώρησης. Δεν μας πέρασε από το πνεύμα να τα αποκλείσουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συστήσει επιχείρηση, όχι μόνο απλώ ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να συστήσει επιχείρηση, αλλά ότι κάθε θηγατρική και υποκατάστημα επιχείρηση έχει συσταθεί από νομικό πρόσωπο, που είναι η μητρική. Επομένω, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να δίδεται αυτή η δυνατότητα για την ηλεκτρονική καταχώρηση. Γιατί τώρα αυτό να είναι πιο δύσκολο στον, στην επαλήθευση του νόμιμου αντιπροσώπου, ενός νομικού προσώπου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πάντα υπάρχει φυσικό πρόσωπο που ορίζεται νόμιμος αντιπρόσωπος ε, ε, νομικού προσώπου. και αυτό καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρό των Εταιριών. Επομένω, οπωσδήποτε στο πεδίο εφαρμογή πρέπει να υπάρχουν τα νομικά πρόσωπα. Μηνύς είναι 36 μέρες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ε, κατά των, της μονομερούς επιβολής ε, άδικων συνθήκων εργασίας από τη δίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένες καμπίνες έχουν, έχουν επιταχθεί, η ε, ελληνική όχι, αλλά σε ένδειξη συμπαράστασης δεν κάνουμε διακοπές εργασίας, ωστόσο δεν δίνουμε παράταση ωραρίου πέραν της προσδιορισμένης ώρας της συνεδρίας. Σας ευχαριστούμε και λυπούμαστε για την τελεπορία. Uh, a member in the Uri Committee, I'm also in the, uh, was also in the Panama Papers Committee and, and right now in the Taxe 3. And I can assure you, we are really fighting that uh, a better registration of the real owner, I mean the one behind all the legal ownership constructions, uh, can be